Uh, good afternoon, everybody. I think we should make a start, even though we're running slightly behind time, because we now have our, our rapporteur here for... Ο εισηγητής μας είναι εδώ για το πρώτο σημείο. Οπότε, επισήμως, να ζητήσω από τους παρόντες συναδέλφους να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Πολύ ωραία. Εγκρίνεται. Απλώς να σας θυμίσω και θα γίνει πληρέστερη ανακοίνωση και πριν τις πληροφορίε όταν έρθουν περισσότεροι συνάδελφοι ότι έχουμε web streaming μετάδοση και από την ε, συνάντηση των συντονιστών ε, την περασμένη εβδομάδα θα ενημερώσω όταν έρθουν περισσότεροι συνάδελφοι. Επίσης έχουμε τα πρακτικά από την ημερίδα για την εσωτερική αγορά που οργάνωσε η ΙΜΚΟΣ Ακρόαση που θα κυκλοφορήσουν στο τέλος της συνεδρίασης. Πάμε λοιπόν στο σημείο που θα καλύψουμε ως 3.30. Πριν ψηφίσουμε στις 3.30 να θυμίσω ότι θα χρειαστείτε τις κάρτες σας για την ηλεκτρονική ψηφοφορία και έχουμε ήδη ξεκινήσει σήμερα τη διαδικασία διαδικασία εξέτασης και υποβολής τροπολογιών τη πρόταση τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερική Αγορά για τη δική τη συνεργασία μέσω του Συστήματο Πληροφόρηση για την Εσωτερική Αγορά, κανονισμό IMI, όπω είναι γνωστό. Ε, ο συγκεκριτή μα είναι ο κύριο Μπίλαν από την ομάδα των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών και έχουμε την κυρία Κολάρη Σαμπίλτ από την. Ε, ω σκιώδη Οι φιλελεύθεροι δεν είναι πολλοί ακόμη, μάλλον θα έρθουν. Αλλά για την ώρα έχουμε μόνο την κυρία Κοράτσα Μπίλτ. Έχουμε και την κυρία Μάριαν Κοράμπεν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα πάρει το λόγο σε λίγο για το ίδιο θέμα. Και επίση υπάρχει και ένα ισχυρό ζήτημα από το Συμβούλιο. Που και εκεί είναι, είναι ευπρόσδεκτη στη συζήτησή μα. Να δώσω λοιπόν τον λόγο στον συγκεκριτή μα, τον κύριο Μπίλαν, για να παρουσιάσει την πρότασή του και τα ζητήματα που έχει εντοπίσει να μας δείξει ποια θα είναι η προσέγγιση του και να μας επιβεβαιώσει και το χρονοδιάγραμμα. Thank you, uh, Mr. Chairman. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να πω ότι είναι πολύ θετική η στάση μου προς την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εντός ολίγου θα σας πω περισσότερα για την πρόταση κανονισμού. Το σύστημα IMI παρουσιάστηκε το 2008 δεκτικά στα κράτη-μέλη ως μια πλατφόρμα πληροφορικής για διοικητική συνεργασία. Πρόκειται για ένα σύστημα διασυνοριακό που θα επιτρέπει τη συνεργασία των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών του ΕΟΧ, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Το σύστημα που ήδη υπάρχει χρησιμοποιείται βάσει της οδηγίας 33 του 2005 για τα επαγγελματικά προσόντα και η οδηγία αυτή 133 συνδυάζεται μάλλον με την 133 οδηγία 33 για τις, εσωτερικές, για τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά. Έχουμε 20 καταχωρήσεις στο σύστημα ημερησίως και Μιλάμε για ένα σύστημα οριζόντια λειτουργία, ένα εργαλείο το οποίο χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή πληροφοριών σε διαφορετικές σε διαφορετικού τομεί, διαφορετικέ θεματολογίε, θα μπορούσε να διευρυνθεί λοιπόν στο μέλλον. Όπω τον τομέα των δικαιωμάτων των ασθενών, όπου υπάρχουν σχετικέ εξελίξει. Θα μπορούσε το σύστημα να χρησιμοποιηθεί για το Solvit ή για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Πρέπει λοιπόν να τονιστεί ότι συνολικά το σύστημα IMI θα έχει πολύ θετικέ συνέπειε για τη λειτουργία τη εσωτερική αγορά. Είναι ένα αξιόλογο εργαλείο για να επιτρέψει την εύρυθμη λειτουργία τη. Να εντοπίσω μερικά ζητήματα για τη λειτουργία του υπάρχοντος συστήματος και για το τι θα θέλαμε να γίνει στο μέλλον εάν ε, επεκταθεί σε νέες θεματικές, σε θεματικούς τομείς. Πρώτον, ο μηχανισμός που αναφέρεται στην ατολική σκέψη 10. Ο μηχανισμός προειδοποίησης. Οι μηχανισμοί αυτοί αναπτύσσονται βάσει συγκεκριμένων συμφώνων. Όμω, ε, θεωρώ ότι ο κανονισμό IMI, λόγω του οριζόντιου χαρακτήρα του, διευκρινίζει ότι η λειτουργία αυτών των μηχανισμών θα πρέπει να ορίζεται λεπτομερώς. Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι ενδιασμοί για τα άρθρα 13 και 14 του κανονισμού επίσης, όπου αναφέρεται η συντήρηση των δεδομένων, η κράτηση των δεδομένων. Ε, δικαιολογείται για 18 μήνες η παρακράτηση των ε, δεδομένων, όμως δεν ξέρω κατά πόσον μπορεί να δικαιολογηθεί πενταετής διάρκεια σε αυτή την περίπτωση. Πρέπει να διευκρινιστεί ποιος θα έχει πρόσβαση στα δεδομένα αυτά και σε ποια νομική βάση στηριζόμενος. Αυτά θα πρέπει να διευκρινιστούν και θα φροντίσω να γίνει αυτό στην έκθεσή μου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να μην διεξαγάγει μελέτη αντικτύπου για τον κανονισμό αυτό και νομίζω ότι αυτό είναι συνετό. Μια τέτοια αποτίμηση θα μπορούσε να συνοδεύει το σχέδιο κανονισμού. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν που θα επεκταθεί το σύστημα, σε κάθε χρονική φάση θα πρέπει να υπάρχει μια σχετική μελέτη. Επίσης μελέτη αντικτύπου για την προστασία δεδομένων θα έπρεπε να συζητήσουμε. διότι το ζήτημα της προστασίας των δεδομένων, εφόσον επεκταθεί και σε άλλες θεματικές περιοχές, σε άλλους θεματικούς τομείς το σύστημα EMI, θα πρέπει να συζητηθεί. Ήδη Είχαμε την πρώτη συνάντηση με τους κοιόδη εισηγητές σε επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου και θα ήθελα και οι υπόλοιπες πολιτικές ομάδες να δείξουν ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο ζήτημα. Γνωρίζω ότι ο χρόνος μας πιέζει, Πρόεδρε. Οπότε θα ήθελα να σας δώσω και το χρονοδιάγραμμα. Σήμερα έχουμε ανταλλαγή απόψεων. Μέχρι τις 16 Ιανουαρίου θα ήθελα να, έχει να, μετα... να αποσταλεί για μετάφραση το σχέδιο έκθεσης. Στις 16 Φεβρουαρίου θα αποφασίσει, θα αποφανθεί η Επιτροπή μας για το σχέδιο έκθεσης. Οι τροπολογίες θα πρέπει να έχουν υποβληθεί ως τις 28 του Φεβρουαρίου στις 12 το μεσημέρι και θα μπορούσαμε να συζητήσουμε τις τροπολογίες στις 21 Μαρτίου και να ψηφίζουμε τον Μάιο. Αυτά από τη δική μου πλευρά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Μπίλαν. Νομίζω ήταν πολύ σαφή η παρουσίασή σα και σωστά δώσατε έμφαση σε κάποια τα ζητήματα που σα απασχολούν. Ξέρω ότι συναντηθήκατε με του και συζητητέ, αλλά είχαμε και μία αποτίμηση από την αρχή που είναι υπεύθυνη για την προστασία των δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Α ακούσουμε λοιπόν τώρα του σκιώδει εισηγητέ. Να ξεκινήσουμε με την κυρία Κοράτσα Μπίλτ, μετά θα ακούσουμε την κυρία Σάλντε Μόζε. Ο κύριο Λόκεγκαρντ είναι επίση σκιώδη εισηγητή. Και η κυρία Ρούιλα φαίνεται να, ότι θέλει το λόγο. Ο κύριο Τρανταφυλλίδη δεν είναι ακόμη εδώ. Ας ακούσουμε την κυρία Κοράτσα Μπίλτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι μεγάλη μου χαρά που μπορώ να ασχοληθώ με την έκθεση αυτή εκ μέρου του ΕΛΚ, διότι θα πρέπει με ένα πολύ πρακτικό τρόπο να αρθούν οι φραγμοί και τα διοικητικά άχθη που βαρύνουν την εσωτερική αγορά που πρέπει να ξεπερνά τα σύνορα. Εδώ θα πρέπει λοιπόν να έχουμε μια δίκαιη, ισότιμη αγορά, ώστε να υπάρχει πραγματικά ελεύθερη κυκλοφορία. Καλωσορίζω την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι νομίζω ότι είναι πραγματικά αξιόλογη. Δημιουργούμε μια, ένα ενιαίο οριζόντιο εργαλείο, προκειμένου να επεκταθεί και να αναπτυχθεί και σε άλλου τομεί, σε βάση τη τεχνική αποτίμηση και να μειωθεί η περιττή γραφειοκρατία, καθώ και να αποφευχθεί η αύξηση του περίπλοκου χαρακτήρα με αυτή την επέκταση. Να πω στον κύριο Μπίλαν ότι έχω την τάση να πιστεύω ότι δεν υπάρχει πραγματική ανάγκη για πλήρη μελέτη δικτύπου. Όλες οι προποθέσει και οι σχετικοί παράγοντε έχουν ληφθεί υπόψη. Εδώ μιλάμε για ενοποίηση υπάρχοντος κειμένου. Δεν είναι πραγματική διεύρυνση. Πιστεύω από νομική άποψη η Επιτροπή έχει κάνει όλα τα δέοντα. Ε, μια μελέτη δικτή που θα προκαλέσει υπερτές καθυστερήσεις και διοικητική εργασία. Εδώ αυτό που θέλουμε να ακούσουμε είναι οι απόψη των ενδιαφερομένων που έχουν ασχοληθεί με το θέμα αυτό σε πρακτικό επίπεδο, περιφερειακό, τοπικό, ξέρουν πώς λειτουργεί το σύστημα και ποιες είναι οι πραγματικές προκλήσεις. Συμφωνώ με τον κύριο Μπίλαν ότι υπάρχει θέμα με το απόρριτο και την προστασία των δεδομένων είναι καθοριστικής σημασίας αυτό, εφόσον θέλουμε την επέκταση του συστήματος. Στο άρθρο 11 θα μπορούσαμε να προτείνουμε το σεβασμό των εθνικών και ευρωπαϊκών κανόνων για την εμπιστευτικότητα και την πρόσβαση στα δεδομένα. Λόγω χάρη για τα έγγραφα. Θα μπορούσε ένα έγγραφο όταν πηγαίνει από μια χώρα στην άλλη να ακολουθείται η νομοθεσία της ε, χώρας ε, παράλληλη αποδοχής. Τώρα για τις κατεξουσιοδότηση πράξεις. Εφόσον επεκταθεί το σύστημα, θα πρέπει να αναθέσουμε στην Επιτροπή να δει τα τεχνικά ζητήματα. Εφόσον υπάρχουν όμω εχέγγυα. Διότι υπάρχουν προτάσει στο κείμενο τη Επιτροπή που είναι πολύ καλά, όπω το δίμηνο για το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, ώστε να αντιδράσουν ότι ετησίω θα πρέπει η Επιτροπή να μα υποβάλει έκθεση, αλλά και άλλε εγγύσει και εχέγγυα θα μπορούσαν να ξέρουμε. Πάντω η καταξιοδότηση πράξη είναι μια λύση. Να ευχαριστήσω λοιπόν τον κύριο Μπίλαν και του υπόλοιπου ε, σκιώδει και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε κυρία Κοράτσα Μπίλτ, κυρία Σάλτερ Μόζε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον, τον ε, εισηγητή για την εργασία που έχει κάνει. Θα μπορέσουν να συζητήσουν το θέμα οι άλλε πολιτικές ομάδες. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι είναι η πρώτη φορά που συμφωνώ με την κυρία Κόρα Ζαμπίλ. Και εγώ προσωπικά θεωρώ ότι είναι πρόταση, σωστή η πρόταση της Επιτροπής και, και από την πλευρά των σοσιαλιστών σε αυτή την πρόταση βλέπουμε τη δυνατότητα να βελτιωθεί η εσωτερική αγορά, να γίνει κάποια πρόοδος. Επίσης να πω ότι κατά την άποψή μας δεν χρειάζεται ίσως να, γίνει να προβλεφθεί μία έκθεση επιπτώσεων. Τη διάταξη που θα έχουμε θα μπορέσει ίσως να μας επιτρέψει να λειτουργήσουμε σωστά. Είχα ρωτήσει μια φορά για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να βελτιωθούν οι διατάξεις που αφορούν την εσωτερική αγορά και η απάντηση που με δόθη ήταν η εξή ότι όλα εξαρτώνται από τον τρόπο με τον οποίο είναι η εφαρμογή του, της νομοθεσίας. Άρα αυτή η πρόταση πάει προς ίσως την κατεύθυνση. Όσον αφορά την προστασία των δεδομένων υπάρχει κάτι, ένα σημείο στο οποίο διαφωνώ, είναι το θέμα των ημερομηνιών. Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει από εκείνου να πάρουν απόφαση. Δεν μπορούμε, δεν μπορούμε να το παρακάμψουμε αυτό με ε, καταστάσεις που θα ρυθμιστούν από εκπροσώπους. Αυτό έχει να κάνει με τη συναπόφαση το θέμα και το καταλαβαίνω ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να σεβαστούμε. Ο κύριος Λόγκαρτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για να συμπληρώσω σε είπε η Δανή συνάδελφος. Νομίζουμε, θεωρούμε μάλλον στην ομάδα Άλντε, ότι είναι ωραία η πρόταση. Καλή. Σημαντικό νομίζω είναι Σαν εκπροσωπώ δεν είναι κυβέρνηση μιλάω, αλλά δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, Το σκεπτικό μας δεν είναι αυτό της κυβέρνησης, αλλά ξέρω ότι η κυβέρνησή μας ενδιαφέρεται το θέμα αυτό να ολοκληρωθεί πολύ γρήγορα κατά το πρώτο εξάμεινο το 2012. Ελπίζω ότι κάτι τέτοιο θα το πετύχουμε. Έχουμε πολλές πιθανότητες. Θα πρέπει να ακολουθήσουμε λοιπόν το ρυθμό που ήδη έχουμε. Και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Κάποιες λεπτομέρειες τώρα. Πιστεύω ότι η πρόσβαση πρέπει να υπάρχει μόνο για την αρχή του IMI και τους χρήστες του. Είναι ένα δικαιτικό εργαλείο, κατά πρώτον. Στο άρθρο 10, παράγραφο 7, θα πρέπει να διευκρινιστεί περαιτέρω ποιοι είναι αυτοί οι ενδιαφερόμενοι που αναφερόνται. Απόψη μου είναι ότι η πρόσβαση για του εξωτερικού ενδιαφερομένους θα πρέπει να επιτρέπεται προκειμένου να υπάρχει και προστασία των πληροφοριών. Επιθυσίες ήθελα να εντυπώσω κάτι στο 18.1, στο άρθρο 18.1. Πιστεύουμε ότι οι κανόνες πρόσβασης για τα δεδομένα θα πρέπει να υπόκεινται στην εθνική νομοθεσία. Ενώ το δίμηνο για τη διαγραφή των ασφαλμένων πληροφοριών μου φαίνεται αρκετά μεγάλο. Δεν χρειάζεται τόσο μεγάλο διάστημα, 60 ημέρες. Δεν δικαιολογείται να σκεφτούμε αν τόσες μέρες χρειάζονται πραγματικά. Να το δούμε. Επιπλέον. Επίση, δεν καταλαβαίνουμε πάρα πολύ γιατί οι τέτοιε χώρε θα έχουν πρόσβαση στα δεδομένα για Ευρωπαίου πολίτε και εταιρείε στο άρθρο 22. Αυτό, κατά την άποψή μου, θα πρέπει να περιοριστεί. Βέβαια αυτά είναι λεπτομέρειες συνολικά. Νομίζω ότι η πρόταση είναι πολύ καλή και θα τη στηρίξουμε. Ελπίζω θα έχουμε μια καλή συνεργασία μεταξύ των σχεδόν. Ευχαριστώ. Thank you very much. Uh, Mrs. Ruler. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ρούλε. Staater bedanken und gleichzeitig entschuldigen, weil ich ja gesagt habe, ich hole noch die Meinung der Stakeholders ein. Das wird aber erst in der Straßburg-Woche klappen und dann werde ich mich auch bei ihm zurückmelden. Äh,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 και όσον αφορά το χρονοδιάγνωμα και πώς θα εξελιχθεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω δεν έχουμε αλλού σκιώδεις. Ο κύριος Φαμπ φαίνεται να θέλει να παρέμβει. Αν υπάρχει κάποιο άλλο, παρακαλώ, κάντε μου νόημα μετά τον κύριο Φαμπ. Και θα ακούσουμε μετά και την παρέμβαση τη Επιτροπή. Κύριε Φαμπ. Vielen Dank, Ich Θα ήθελα να πω ότι χαίρομαι για την συμφωνία που υπάρχει όσον αφορά αυτή την πρόταση. Θεωρώ ότι για την εσωτερική αγορά έχουμε τα σημαντικά εδώ μέσα για να μπορέσουμε να ε, εφαρμόσουμε την οδηγία αλλά και άλλες οδηγίες στο μέλλον. Είναι πραγματικά ένα μέσον το οποίο θα μας επιτρέψει να περάσουμε στη βράξη. αυτό το σύστημα λειτουργεί καλά και θα πρέπει μάλλον να λειτουργήσει ξανά, διότι από αυτό θα εξαρτηθεί αν θα ικανοποιηθούν τα διάφορα μέρη, χώρες μέλη, αυτοί τους οποίους αφορά και για όλους όσοι ενδιαφέρονται ε, επαγγελματικά. Θα ήθελα όμως να πω ότι κατ' εμέ υπάρχουν κάποιες πτυχές οι οποίες έχουν να κάνουν με περιπτώσεις, ποιες θα είναι οι περιπτώσεις στις οποίες θα αφορά το σύστημα. Η Επιτροπή φυσικά θεωρεί καταρχήν ότι το σύστημα λειτουργεί σωστά. Εγώ θεωρώ όμως ότι δεν έχουμε πολύ ικανοποιητική ε, κατάσταση. Υπάρχουν πράγματα τα οποία θα πρέπει να ρυθμιστούν. Υπάρχουν ειδικέ περιπτώσεις όπου βλέπουμε ότι έχουμε ελλείψεις για το όσον αφορά την ε, λειτουργία συστικά με τις μεταφράσεις. Υπάρχουν δηλαδή τα προβλήματα που αφορούν καθαρά το γλωσσικό επίπεδο, το πέρασμα στη μετάφραση και θα ήθελα να πω στους συναδέλφους μου ότι μέχρι στιγμής έχουμε μια περιορισμένη χρήση περιπτώσεων μέσω αυτού του συστήματος. Ε, όσον αφορά την αναγνώριση των ε, ε, επαγγελματικών προσόντων Φερπίν. Γι' αυτό θα πρέπει να κοιτάξουμε πώς μπορούμε να δοκιμάσουμε αυτό το σύστημα, να δούμε πώς αντιδρά όταν έχουμε να κάνουμε ε, μεγάλο, αριθμό περιπτώσεων. Έχουμε τώρα να κάνουμε μια περίπτωση που αφορά τη διαδικασία συνεργασίας. Ε, θα πρέπει η Επιτροπή να έχει κάποιες αρμοδιότητες δεν θα είναι, θα είναι δυνατόν ή δεν κάποια άτομα να μπορέσουν να δεχθούν προτάσεις. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω άλλος να θέλει να παρέμβει. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στον κύριο Μπίλαν για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση σε λίγο. Αλλά προηγουμένω θα ήθελα η εκπρόσωπο τη Επιτροπή, την οποία καλωσορίζω, να μα παρουσιάσει τι απόψει τη Επιτροπή και να σχολιάσει όσα είπαν οι συνάδελφοι βουλευτέ. Ευχαριστώ κύριε Χάρμπορ. Είναι χαρή, χαρά μου που ακούω τόσο θετικέ αντιδράσει για τον ε, κανονισμό IMI. Βεβαίω έχουμε ξαναέρθει στην Επιτροπή σα για να εξηγήσουμε τι προγραμματίζουμε για την επέκταση του IMI σε, σε άλλους τομείς θεματικούς. Ο κανονισμός αυτός είπαμε ότι είναι απαραίτητος προκειμένου να μπορέσουμε να επεκτείνουμε το σύστημα σε άλλους πολιτικούς τομείς. Αντιδρώντα τώρα στα όσα είπε ο κύριο Μπίλαν για την μελέτη δικτύπου που δεν έχει γίνει, το εξετάσαμε προσεκτικά βεβαίω. Όμω, όπω είπαν και κάποιοι από του ομιλητέ, ο κανονισμό αυτό απλώ ενωπεί ένα σύστημα το οποίο ήδη λειτουργεί κανονικά. Εδραιώνει του κανόνε προστασία των δεδομένων που ήδη εφαρμόζονται. Απόψη μα λοιπόν ήταν ότι ο κανονισμό αυτό καθεαυτό δεν προκαλεί πρόσθετο κόστο και η εξαγωγή μελέτης αντικτύπου δεν είναι απαραίτητη. Βέβαια, συνειδητοποιούμε ότι εφόσον αποφασίσουμε να επεκτείνουμε το σύστημα σε άλλους πολιτικούς τομείς, θα χρειαστεί μελέτη αντικτύπου. Αυτή θα είναι μέρος της τομεακής νομοθεσίας που την απαιτεί. Κάτι άλλο για την περίοδο κράτησης των δεδομένων. Οι 18 μήνες είναι καθοριστική σημασία για να διασφαλίσουμε ότι οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επεξεργαστούν αιτήσει από ετούντο λόγου χάρη που θέλουν να μάθουν τι έγινε με του φακέλου του IMI. Επίση υπάρχει και μια περίοδο κράτηση πενταετία για κάποια δεδομένα. Δεδομένα τα οποία θα ε, είναι αποκλεισμένα. Δεν θα μπορεί κανεί να έχει πρόσβαση σε αυτά. Εάν οι αρμόδιε αρχέ τα χρειάζονται μετά από αίτηση των ε, ενδιαφερομένων, θα πρέπει να υπάρξει τεχνική παρέμβαση για να αποσπαστούν. Η πεντέτης. λοιπόν ε, περίοδος είναι μια εγγύηση ώστε να εξασφαλιστεί η άσκηση του δικαιώματος των ετούντων να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα τους. Το πρώτο πραγματικό παράδειγμα που θα αντιμετωπίσουμε σε σχέση με, την, με τους εξωτερικούς ενδιαφερομένους είναι με την ε, συμπερίληψη τη εφαρμογή Solvit στο σύστημα IMI, διότι η εφαρμογή αυτή ήδη επιτρέπει στου ε, πολίτε και τι εταιρείε να υποβάλουν ε, online επιγραμμική ε, υποβολή, να υποβάλουν μάλλον στο διαδίκτυο τα παραπονά του. Αυτό θα ολοκληρωθεί στο σύστημα AMI. Σε ό,τι αφορά τι τρίτε χώρε, υπάρχουν συγκεκριμένε προποθέσει υπό τι οποίε θα είναι δυνατόν να διασυνδεθούν οι αρμόδιες αρχές των ε, τρίτων χωρών στο σύστημα IMI. Μεταξύ αυτών είναι να υπάρχει μελέτη καταλληλότητας για την ε, προστασία των προσωπικών δεδομένων στις τρίτες αυτές χώρες. Επίσης, σημαντικό είναι τρίτες χώρες να έχουν εγκρίνει τουλάχιστον ένα νομοθέτημα της ε, Ένωσης μέρος του κανονισμού IMI. Λόγου χάρη, σκεφτόμασταν την συμφωνία που πρόσφατα πετεύχθη με την Ελβετία για την εφαρμογή του σε σχέση με την οδηγία της, ε, των επαγγελματικών προσόντων. Θα ήταν πρακτικό σε αυτή την περίπτωση αν οι αρμόδιε αρχέ τη Ελβετία μπορούσαν να ανταλλάσσουν αρχέ με αυτέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμω το άρθρο αυτό ουσιαστικά απλώ δίνει τη δυνατότητα. Δεν καθορίζει ποιε χώρε τελικώ θα αποτελέσουν μέρο του συστήματο. Σε ό,τι αφορά τι απόψει των ενδιαφερομένων εδώ, Μα ενδιαφέρει πολύ να έχουμε την απόκριση των πραγματικών χρηστών του συστήματο και το τι πραγματικά πιστεύουν για το σύστημα. Εάν το θέλει η Επιτροπή σα, μπορούμε να δώσουμε και στατιστικά στοιχεία για τι πιο πρόσφατε έρευνε μα για το θέμα αυτό. Θα μπορούσατε να δείτε τι σκέφτονται οι πραγματικοί χρήστε για το σύστημα EMI. Επίση, μα ενδιαφέρουν τεχνικέ βελτιώσει του συστήματο να ολοκληρωθούν ώστε να γίνει πιο φιλικό προ το χρήστη από ό,τι είναι σήμερα. Ω προ το ζήτημα το γλωσσικό, Πέρυσι είχαμε ένα πρόβλημα με τα μηχανήματα μετάφρασης ε, του IMI, αλλά προσπαθούμε να το διορθώσουμε όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Ελπίζουμε και έχουμε βάσιμες ελπίδες ότι το προηγούμενο μηχανικό μεταφραστικό σύστημα θα έχει ε, διορθωθεί ως τον ερχόμενο Μάρτιο ή Απρίλιο. Σε ό,τι αφορά τον όγκο ετήσεων του συστήματος IMI, το σύστημα έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να χειρίζεται 100.000 αιτήσει περίπου ετησίω. Ήδη ο όγκο αυτό είναι περιορισμένο. Νομίζω λοιπόν ότι δεν θα υπάρχουν προβλήματα ως προς τον, ε, την κλίμακα ενώ οποία λειτουργεί το σύστημα άμεσα. Και ως προς την οδηγία για τα επαγγελματικά προσόντα και την πρόταση που επίκειται, Υπάρχει εδώ ένα ε, σημαντικότερο ρόλο που θα διαδραματίσει το σύστημα IMI. Αν σκεφτείτε πώ ήδη λειτουργεί το σύστημα, νομίζουμε ότι εύκολα θα μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε χωρί προβλήματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Να θυμίσω σε όλου, δίνοντα έμφαση σε αυτό που είπατε στην αρχή τη παρέμβασή σα, ότι η πρόταση αυτή είναι πολύ σημαντική ως ένα μέρος της ε, πράξης της ενιαίας αγοράς, ένα από τα 12 στοιχεία της πρότασης αυτής. Θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο. Θέλουμε λοιπόν ε, να το αντιμετωπίσουμε το ζήτημα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και με επιτυχία. Να ξαναδώσω το λόγο στον εισηγητή μα, τον κύριο Μπίλαν, για να με ανακεφαλαιώσω όσα ήδη υπόθηκαν ενδεχομένω. Έχετε ήδη καθορίσει το χρονοδιάγραμμα. Μπορεί να έχετε και κάποια πρόσθετη παρατήρηση πριν κλείσουμε τη συζήτηση για το σημείο αυτό. Κύριε Μπίλαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Γνωρίζω ότι θα πρέπει άμεσα να ξεκινήσουμε την ε, ψηφοφορία. Ευχαριστώ τους σκιώδεις εισηγητές για τα σχόλια που κάνα και για την καλή συνεργασία που είχα μαζί τους. Σίγουρα θα μπορέσουμε να ξανασυναντηθούμε πριν να διεκπαιρωθούν όλες αυτές οι προθεσμίες. Επίσης, να ευχαριστήσω την Επιτροπή για, τη λεπτομερή, για το λεπτομερή σχολιασμό και για όλες τις ε, αμφισβητούμενες ε, πτυχές αυτού, αυτής εκθέσεως. Ελπίζω να εγκριθεί αυτή η έκθεση για να αποτελέσει μια επιτυχία για τη Δανέζικη Προεδρία. Ευχαριστώ πολύ. Well, Σας ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά προσβλέπουμε στη συζήτηση της έκθεσής σας μετά τα Χριστούγεννα και θα δούμε τι συνέχεια θα δοθεί. Λοιπόν, ας περάσουμε τώρα στην ώρα των ψηφοφοριών. Πριν το κάνω αυτό, μια που έχουμε αρκετά μέλη παρόντα, Make the... Σας κάνω μερικές ανακοινώσεις. Συνεδρίασαν συντονιστές την περασμένη εβδομάδα. Πρώτο, ανάθεση εκθέσεων ε, προς ενημέρωσή σας πρόταση για κανονισμό Συμβουλίου και Κοινοβουλίου για το πρόγραμμα κατά 2014-2020. φιλελεύθερη το αναλαμβάνουν αυτό. Άλλη πρόταση για την προσαρμογή και την ευθυγράμμιση διαφόρων προϊόντων marketing θεωρείται τεχνική έκθεση να λαμβάνει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Δύο εκθέσεις που συνδέονται εναλλακτική επίλυση διαφορών και διακανονισμό και επίγραμμα. Και ο κύριος Γκρέχ θα κάνει την πρώτη από τους σοσιαλιστές και τη δεύτερη ε, από το ΕΛΚ, μία συνάδελφος. Αυτές ήταν οι βασικές ε, αποφάσεις. Θα τις βρείτε και στην ιστοσελίδα συζητήσαμε και για τις αποστολές του 2012. Κάτι άλλο σημαντικό σε σχέση με τις μοτοσυκλέτες και θα έρθω στη συνέχεια σε αυτό. Οι συντονιστές επιβεβαίωσαν και τυπικά το αίτημά του για να δοθεί ειδική προσοχή και εξέταση μια μελέτη αντικτύπου και σκοπιμότητας για τις τροπολογίες της Επιτροπής μας που θα επιβαρύνουν και οικονομικά την πρόταση. Την έκθεση αυτή θα την εξετάσουμε και στη συνέχεια. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει τελειώσει εδώ. Πριν ολοκληρωθεί όμως η νομοθετική προσπάθεια θα ενημερωθείτε και θα συζητήσουμε και για αυτό το θέμα της οικονομικής επιβάρησης. Ωραία. Τι άλλο ήθελα να σας πω. Σήμερα το πρωί συνεδρίασε το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας για να συζητήσει τα αποτελέσματα του Φόρουμ Αγοράς. Γνωρίζω ότι πολλοί από εσάς ήσασταν παρόντες το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας ενέκρινε ένα ψήφισμα εκτενέστατο που ε, σχολιάζει και λεπτομέρειες και συμπεράσματα της δήλωσης του φόρου και ως Επιτροπή θα ήθελα να τα συζητήσουμε για να τα γνωρίζετε αλλά και δημόσια. Το Συμβούλιο λέγει ότι καταρχάς καλωσορίζει πάρα πολύ καλά τη ε, δήλωση αυτή και χαίρεται για τη δέσμευση όλων των ενεχομένων τόσο πολλών και παραθέτω ε, εκτιμά την προσπάθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την καλή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που κατέστησαν δυνατή την εκδήλωση αυτού του ε, άνευ ε, προηγουμένου γεγονότος. και αυτό θα μπει στην ιστοσελίδα και θα κυκλοφορήσει για τα μέλη. Ήταν μια διοργάνωση που έγινε πρώτη φορά. Καλώς. Λοιπόν, προχωρούμε στις ψηφοφορίες μας και με πρώτο θέμα έγκριση γεωργικών και δασικών οχημάτων. Ο εισηγητής είναι εδώ, είναι παρόν ο κύριο Παντσέρη. You are in charge of the Uh, Δυστυχώ ο κύριο Πανσέρη κολλείεται και απουσιάζει. Τον αναλαμβάνει η κυρία Βερνιό. Θα τη δώσω αμέσω στο λόγο εξ του εισηγητού και πριν ψηφίσουμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα εκ μέρου του Αντώνιου Παντσέρη να ζητήσω συγγνώμη. Έμεινε ε, στην Ιταλία σήμερα, αλλά θα γίνει η ψηφοφορία μου είπε κάποια πράγματα, ότι ευχαριστεί όλους τους σιώδης για τη συνεργασία τους σε ένα θέμα το οποίο είναι πολύ τεχνικής φύσεως σε σχέση για τα θέματα γεωργικών και δασικών οχημάτων. Ε, υπάρχουν οι τροπολογίες οι οποίες αγγίζουν τα πιο ευαίσθητα σημεία και κυρίως το κεφάλαιο 16, δηλαδή την πρόσβαση στις για τις πληροφορίες σε σχέση με την επισκευές των οχημάτων. Ε, ε, επίσης το θέμα των αποκλεισμών κάποιων οχημάτων, έχουμε τον κανονισμό το οποίο θα πρέπει να εγκριθεί από την Επιτροπή την Ευρωπαϊκή και το θέμα των οχημάτων για και φυσικά για τις ε, διαπραγματεύσεις που έχουν γίνει μέχρι τις τελευταίες μέρες έχουμε καταλήξει σε πέντε συμβαστικές τροπολογίες οι οποίες ε, καλύπτουν όλα τα βέστα σημεία της εκθέσεως και όπου επιτεύχθη η συμφωνία ανάμεσα στις πολιτικές ομάδες. Μόνο η ερώτηση που έχει να κάνει με τα ε, οχήματα τα οποία είναι για όλους τους χώρους, εκεί υπάρχει μια επιφύλαξη Υπάρχει αυτή η κατηγορία λοιπόν η οποία δεν έχει συμπεριληφθεί σε, αυτήν, αυτό το κανονισμό. Και τη στιγμή που θα υπάρχει και μια μελέτη για τις επιπτώσεις θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε στις ομάδες μας οριζοντίως πριν να περάσει η ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Ξανά λοιπόν ε, να ευχαριστήσουμε, ευχαριστήσω από μέρους ε, τους και να περάσουμε στην ψηφοφορία. Καλώς. Ευχαριστώ. Και τους υπόλοιπους εισηγητές ε, εξ ονόματος θα πρέπει να ευχαριστήσουμε. Καλωσορίζω και τον Φιλίψα από τη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων ε, που μας ε, επικουρεί σε αυτό το σημαντικό και περίπλοκο θέμα. Ψηφίζουμε. Οι σκιώδεις συγητές συμφώνησαν ότι μπορούμε να ψηφίσουμε πολλές τροπολογίες μαζί, on block όπως συνηθίζω να το λέμε. Θα ψηφίσουμε αργά για να καταλαβαίνουμε όλοι τι ψηφίζουμε. Συμφωνήσαν οι ε, πολιτικέ ομάδες, συμφωνήσαμε. Νομίζω υπάρχει και μια προφορική τροπολογία. Λοιπόν, κάντε λίγη υπομονή και να μην συμπαθάτε. Θα προχωρήσουμε αργά και όπου ε, χρειάζεται θα γίνεται ηλεκτρονική ψηφοφορία έλεγχος, αλλά κατά κανόνα δυνατά χειρός Θέλει κανείς και να μιλήσει, όχι. Λοιπόν, ψηφίζουμε. Έχουμε μια ε, μαζική ψηφοφορία 1, 15, 16 στο άρθρο 1, 17, 18, 19 και 307 στο άρθρο 2. Όλα αυτά μαζί. Ψήφι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Επόμενες δύο που έχουν αποσυρθεί. Και τώρα ψηφίζουμε. Δύο ταυτόσημες για το άρθρο 2 παράγραφος 2. 3, 10, 3, 11 ψήφι υπέρ κατά εγκρίνονται. Άλλο μπλοκ τώρα. Τροπολογία 20, 21, 312, 313, 22 υπέρ όλων αυτών κατά εγκρίνονται επίσης. Τώρα 314 και 316 ψήφι υπέρ. Ταυτόσιμες αυτή κατά εγκρίνεται. 315 έχει αποσυρθεί. Και τώρα μεγάλο μπλοκ και πάλι ε, δούμε 317-318, ε, συγγνώμη, 23-24-25, 319 και 320 έχουν αποσυρθεί, 26 και 27 δεν τα ψηφίζουμε, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 και 34, λέει ο πρόεδρος. Μέχρι εκεί είναι το μπλοκ αυτό, υπέρ, κατά εγκρίνονται όλα αυτά. Τώρα ψηφοφορία χωριστή για την 35 ψήφι υπέρ της τροπολογίας 35 κατά. Εγκρίνεται με μεγάλη άνεση. Άλλο μπλοκ τώρα, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 δεν τις ψηφίζουμε. 42, συγγνώμη, 43, 44, 45, 46, 47 και 48 και 49. Μαζί όλες αυτές, υπέρ. Κατά. Όλες αυτές συγκρίνονται. Άρθρο 3, παράγραφος 1. 321 είναι η τροπολογία χωριστή. Αφορά τη μέγιστη ταχύτητα. Ψηφίζουμε το σύνολο του κειμένου χωρίς αυτό το τμήμα υπέρ. Α, εδώ μάλλον χρειάζεται ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται για το πρώτο τμήμα αυτό. Πέρας. Ψηφίζουμε την προφορική τροπολογία για τα 40 χιλιόμετρα. Ψηφίζουμε παρακαλώ για τα 40 χιλιόμετρα. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται στα 60 χιλιόμετρα ψηφίζουμε τώρα ε, άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται σαφώς 50 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τι έχουμε τώρα, η επόμενη καταπίπτει. Right. Okay. So, we, we then on Άρα ψηφίζουμε την 323 τώρα. Η εισηγητής είναι κατά υπέρ κατά Α, Α, άλλα είναι αυτά τα οχήματα, χωριστή ψηφοφόρια. Είναι τα side by side, οχήματα αναψυχής εκτός δρόμου. Το πρώτο τμήμα είναι όλο το κείμενο, χωρίς τις λέξεις. Με έχει ταχύτητα κάνει θειασμό 60 χιλιόμετρα, ψήφι υπέρ. Α, ηλεκτρονικά μάλλον θα γίνει αυτό. Γιατί 321 το πρώτο τμήμα ψηφίζουμε λοιπόν τώρα ηλεκτρονικά το τμήμα αυτό. Πέρας. Απορριπτείται σαφώς. Καταπίπτουν οι υπόλοιπες τροπολογίες. Um... So, we now put to vote the next block. Επόμενο μπλοκ, 51, 52, 53 και 54. Υπέρ, είναι του σύγητου. Κατά εγκρίνονται. Η 55 δεν ψηφίζεται. Τώρα έχουμε χωριστές ψηφοφορίες. 324. Άρχισε η ψηφοφορία. The vote is closed. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 325. Um, the vote is Άρχεται η ψηφοφορία για την 325. Πέρας. Εγκρίνεται και αυτή. Η 326. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Επίσης εγκρίνεται. 327. Υπέ. Α, μάλλον έρθει η ψηφοφορία, συγγνώμη, ηλεκτρονικά. Πέρασε. Εγκρίνεται επίσης. 3.31 θα τα δούμε αργότερα αυτά. 3.38 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Θα σας παρακαλούσα να επιταχύνετε λίγο Τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 329. Ε, Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζεται λίγο πιο γρήγορα, λέει ο πρόεδρος. Πέρας. Εγκρίνεται και αυτή. 331 καταπίπτει. Και 56 και 30 δεν τις ψηφίζουμε. Επόμενο σύνολο. Είναι η τροπολογίες του κυρίου πανσερι 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66. 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84. Ουφ, μέχρι εκεί. Μεγάλη δέσμη τροπολογιών ψήφι υπέρ του εισηγητού κατά αποχές εγκρίνονται. Και τώρα ψηφίζουμε χωριστά την 332 του κυρίου Παντζέρη. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 85 καταπίπτει και πάμε τώρα στο επόμενο σύνολο. 86, 87, 88, 89. Οι, δύο, οι υπόλοιπες έχουν αποσυρθεί και μετά 90 έως και 94. Αυτές όλες ψηφίζουμε μαζί. Ψήφι κατά εγκρίνονται όλες αυτές. Πάμε τώρα στη συμβαστική τροπολογία παριθμών 1. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα 96. Σε άλλο μπλοκ είναι αυτή τώρα. 97, 340, 98, 339, 99, 100, 341, 101, 342, 102, 103, 109, 104, 344, 105 μέχρι και... δεν μην σας τις διαβάζω όλες. Θα σας πω σελίδα τώρα. Δεν ξέρω βέβαια αν έχουμε όλοι τον ίδιο κατάλογο ψηφοφορία. Είναι όλες οι τροπολογίες για το άρθρο 8, 9, 10, 11, 12, 13... Τεχνικές 14, 15, 16 άρθρα είναι αυτά που σας λέγω τώρα, 17, 18, 19, 20, 21, 23 και 193 στο άρθρο 24. Όλα αυτά με παρακολουθείτε μέχρι εδώ. Ψηφίπερ. Κατά. Εγκρίνονται. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Πανσέρη. Έχει εργαστεί πολύ σκληρά σε αυτό το θέμα. 3.48 τώρα. Ψήφι υπέρ. Uh, well, I think we'll open the on this. 348. Νομίζω χρειάζεται ηλεκτρονική επαλήθευση για την 348, παρακαλώ. Πέρασε. Εγκρίνεται. Τώρα, άλλη ενότητα. Για το υπόλοιπο άρθρο 24, 25, Ε, αλλαγή του τίτλου 203, άρθρο 26, άρθρο 27, 28, άρθρο 29 και άρθρο 30. Ε, τροπολογία 227, η πρώτη μόνο. Ψήφι υπέρ. Όλα αυτά τα τροπολογία κατά εγκρίνονται. 228 το ψήφι Κατά εγκρίνεται σαφώς. Και τώρα άλλο μπλοκ. Από την 2.30, 2.31, άρθρο 31, 32, 33, 34, κεφάλαιο 12 τίτλος, ψήφι υπέρ, μέχρι εκεί και την 2.37 κατά εγκρίνονται. Και τώρα, η τροπολογία 3.54, εδώ με προφορική, παρακαλώ, του κυρίου Μάντερς, όπου προτείνει να παληφθεί το δεύτερο τμήμα του άρθρου 35β. Συμφωνούν οι σχεδόν ηγητές καταρχήν το γνωρίζουν. Ναι, είναι τμήμα του συμβιβασμού. Θα το αποσύρω, λέει ο κύριος Μάντερς, και θα ψηφίσουμε μόνο το πρώτο τμήμα. Συμφωνείτε όλοι οι σχεδόν μάλιστα. Ωραία. Το ψηφίζουμε λοιπόν. 354 με την προφορική τροπολογία του κυρίου Μάντερς. Ψήφι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται σαφώς. Ωραία. Άλλο μπλοκ τώρα. Άρθρο 36, 38 και άρθρο 44. Η τροπολογία 248. Μέχρι εκεί. Ψήφι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται σαφώς. 249 του εισηγητή αρχίζει τώρα η ψηφοφορία ηλεκτρονική για τη 249. Πέρας. Απορρίπτεται. Οπότε και θα περάσουμε στην 356-357 με προφορική τροπολογία, όπως βλέπετε στον κατάλογο ψηφοφορίας σας. Ψήφι πέρα. Κατά, εγκρίνεται. καταπίπτουν αν δεν απατώμε 356-357. Πάμε συμβαστική 2 ψήφι πέ. Κατά εγκρίνεται. Και τώρα συνεχίζουμε. με τη 411 γιατί όλες οι προηγούμενες καλύπτονται από τη συμβαστική 411 στο άρθρο 50 ψήφι πέ κατά εγκρίνεται Άλλο μπλοκ τώρα. Τροπολογίες για το υπόλοιπο άρθρο 50 και 51 και 53 και 54, 55, 56, 57 άρθρα όλα αυτά. 58, 59, 60, 61 και μέχρι το συμβιβασμό υπαριθμών 3. Όλες αυτές τις τροπολογίες ψήφι υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 3. Ψήφι Κατά. Εγκρίνεται σαφώ. Στο άρθρο 62 όλες οι τροπολογίες. είπε. Κατά. Εγκρίνονται και οι τέσσερις τροπολογίες. 292 του κύριου Πανζέρη στο άρθρο 63 ψήφιπε. 292. Α, όχι, ηλεκτρονικά ψηφίζουμε την τροπολογία 292. Πέρας. Απορρίψετε. Τώρα πάμε στη συμβαστική υπαριθμών 4 ψήφι Κατά. Εγκρίνεται σαφώ Και ακολουθεί η 2.94. Α, είμαστε στις ιδεολογικές σκέψεις τώρα. 2.94 και άρθρα 3 και 4. Μαζί όλα αυτά. Ψήφι Εγκρίνεται. 295 ως προσθήκη. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Κάποιες τεχνικές ακολουθούν που δεν ψηφίζονται. Η επόμενη που ψηφίζουμε είναι η 296. Αρχίζει η ηλεκτρονική ψηφοφορία για τη 296. Πέρασε. Απορρίπτεται. 8 και 9 δεν την ψηφίζουμε. 2,97 7 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 2,98 σφαπ. υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 2,99 και 300 υπέρ. Νομίζω θα χρειαστεί ηλεκτρονική ψηφοφορία γι' αυτό. 2,99 και 300 μαζί. Άρχεται η Πέρας. Απορρίπτεται. Vote. Ε, ισοπαλία. 301 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Η τροπολογία 10. 11, 12, 13, 306 και 14 υπέρ κατά εγκρίνεται και το τελευταίο αυτό σύνολο τροπολογιών. Οριστική τελική ψηφοφορία ονομαστικά αρχίζει τώρα για την πρόταση όπως τροποποιήθηκε. Παρακαλώ επιταχύνετε την ψηφοφορία σας. Ψηφίσατε όλοι γρήγορα. 31 κάρτες έχουμε και ποιος καθυστερεί 30 είχαν ψηφίσει. Πέρας τώρα ψηφίσατε όλοι. 31 υπέρ, κανείς κατά. Εγκρίνονται λοιπόν οι τροπολογίες. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Πανσέρη και το χειροκροτούμε παρότι απουσιάζει. Σας ευχαριστούμε. Κύριε Πανσέρη, εν τη απουσία σας που ετοιμάστε τόσο καλά ε, την ψηφοφορία και είμαι βέβαιος ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ε, σημειώσει με προσοχή τις λεπτομέρειες και σε ό,τι αφορά τη μελλοντική συζήτηση με το Συμβούλιο. Βλέπω ότι ο εκπρόσωπος της Κομισιόν που συνεργάστηκε στενά με τον εισηγητή νεύει καταφατικά. Επόμενη έκθεση του κυρίου Βαντεκάμπ. Για την έγκριση και εποπτεία της αγοράς δίκυκλων, κύκλων οχημάτων και τετρακύκλων. I haven't got the version. It should be there. Okay. Right. Uh, yes, there it is. So, we approve on the report of Mr. Van der Kamp. Περνάμε στην έκθεση Van der Kamp. Νόμιζα κύριε Σακητάτο θα κατέβετε πιο κάτω. Πρόεδρε, προσπάθησα, αλλά η κάρτα δεν λειτουργεί. Αν εσείς αλλάξετε θέση... Ίσως να μπορεί ένας τεχνικός να το διορθώσει. to introduce the vote. Κάντε μας μια εισαγωγή, εισήγηση για την πληροφορία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πολύ ωραία ήταν η νομοθετική διαδικασία που ζήσαμε με πολλές συνεδριάσεις ε, και πολλούς ενδιαφερομένους και ενεχομένους. Ουσιαστικά τρία είναι τα μεγάλα υποκεφάλαια της έκθεσης. Το πρώτο είναι οι δυνατότητες και ε, τι μπορεί να κάνει δηλαδή και τι δεν μπορεί να κάνει η βιομηχανία μότο ποδηλάτων, μότο και άλλων οχημάτων που είναι πάνω από 100. Ε, οι εταιρείε αυτές. Το δεύτερο είναι η βιωσιμότητα και η αηφορία και ε, με την πρόταση αυτή οι εκπομπές των δικύκλων θα μειωθούν σημαντικά στην Ευρώπη και κυρίως στις αστικές ε, περιοχές. Αυτό είναι κάτι πολύ ωραίο και σημαντικό. Και το τρίτο κεφάλαιο είναι η ασφάλεια των δικύκλων. Κυρίως τα συστήματα τροχοπέδησης συγκέντρωσαν την προσοχή μας ε, το τελευταίο διάστημα. Δεν το έχουμε λύσει ακριβώς για να είμαι αυτό, αλλά προχωρούν οι συνομιλίες. Για τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις ηγητές για την εντατική του συνεργασία, αλλά και τη γραμματεία της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Καταναλωτών και πάντα μας καθησυχάζει το γεγονός ότι η ε, Κομισιόν και ε, το Συμβούλιο ασχολούνται με τα θέματα αυτά και τα παρακολουθούν. Και επίσης είναι και μεγάλη πρόκληση να έχει κανείς και γιατί κάποιον που είναι πρόεδρος της Επιτροπής του. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Βαντασφαντή. Μόνο και για τα ρημαρκούμενα οχήματα και τα μηχανοκίνητα. Εξηγητής. Ε, νομίζω εδώ είναι πολλοί εκείνοι που μας ακούν από το διαδίκτυο την ενδιαφέροντα για το θέμα αυτό. Να πω λοιπόν ότι κάτι που μου ζήτησαν οι σχεδόν συζητητέ είναι ότι ένα από του τομεί που προτείνουν να προβλεφθούν στοιχεία για την ασφάλεια και τις εκπομπές είναι ε, να δούμε τι επιρροή θα έχει μια μελέτη αντικτύπου στο κόστος και το χρόνο ισχύως θέσης ισχύ της οδηγίας. Και επίσης τι θα γίνει με τα συστήματα τροχοπέδησης και τα ειδικά μηχανήματα. Μετά την ψηφοφορία σήμερα βέβαια θα ξέρουμε καλύτερα, γιατί σήμερα θα επικεντρωθούμε κυρίως στις εκατοντάδες τροπολογίες που έχουμε. Πολλοί νομίζω λάβατε ηλεκτρονικά μηνύματα από ανθρώπους που ρωτάνε γιατί ψηφίζουμε πριν δούμε τα αποτελέσματα της μελέτης αντικτύπου. Ο εισηγητή όμω ξέρει πολύ καλά ότι θα δούμε τα πορίσματα τη μελέτη αντικτύπου πριν ψηφίσουμε στην Ολομέλεια και σήμερα μετά την ψηφοφορία θα έχει συζητήσει με το Συμβούλιο για το πώ προχωρούν οι διαπραγματεύσει μα ε, κατά για το θέμα αυτό. Πάντω θα δούμε τα πιο λεπτομερή ζητήματα σήμερα. Κύριε Μάντερ, ναι, για, το, για την επιστολή που θα απευθύνει η δική μα Επιτροπή στην Επιτροπή Μεταφορών. Είναι πολύ σημαντικά τα μοτοποδήλατα αλλά ίσω ακόμη πιο σημαντικό είναι το τι θέλουν οι οδηγοί. Ναι, υπήρξαν πολλέ τροπολογίε που δεν είχαν να κάνουν με την τεχνική διάσταση τη οδηγία. Αυτό μα προκάλεσε κάποιε ανησυχίε. Σκεφτήκαμε λοιπόν ότι ο καλύτερο τρόπο ήταν να αποστείλουμε επιστολή στου συναδέλφου τη Επιτροπή Μεταφορών. Και πολλοί απάντησαν ότι τα δεσμεύματα αυτά διαθετούνται σε 100 μελών. Δεν χρειάζεται ακόμα η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ο εισηγητής μας και ο κύριος Μάντες ως σκεωδής θα ετοιμάσουν λοιπόν σχετική επιστολή που θα εμφανιστεί και στον ιστοτοπό μα. σας. προχωρήσουμε με την ψηφοφορία. Ξεκινούμε με το άρθρο 82. Τροπολογία 60. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Άρθρο 2. Τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 11. Υπέρ κατά εγκρίνεται. Συνολικά 106-110 της κυρίας Ρούιλε υπέρ κατά εγκρίνεται. 13 υπέρ κατά εγκρίνεται. 112 υπέρ κατά εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά εγκρίνεται. 15 εδώ έχουμε τα ψηφοφορία που ζητήθηκε από την Άλντε. Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, σαφώς εγκρίνεται. 16 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 17 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Η 8 εκπληκτή. 18 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η 7 της Επιτροπής Μεταφορών εκπίπτει. 218 το ίδιο. Η 63 έχει αποσυρθεί. Η 219 εγκρίνεται επειδή εγκρίθηκε 18. Και πηγαίνουμε τώρα στη συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Χωρίς αμφιβολία. Περνάμε τώρα στο σύνολο 113 και 114. Συμβαστική τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική λοιπόν 1. Και μετά 20, 21 και 22. Ψηφίζουμε συνολικά υπέρ. Κατά. Εγκρίνονται. Τώρα 23 και 25. Υπέρ κατά εγκρίνονται. 26 υπέρ κατά εγκρίνεται. 87 27 μάλλον συγγνώμη. 119 ε, υπέρ κατά απορρίπτεται. 120 υπέρ κατά απορρίπτεται. 31 υπέρ κατά εγκρίνεται. 121 υπέρ κατά εγκρίνεται και 32 13 στην Επιτροπή Μεταφορών υπέρ κατά εγκρίνεται. 33 και 14 της Επιτροπής Μεταφορών υπέρ κατά εγκρίνονται. 124 υπέρ κατά εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 3. Τι έγινε. Κατέχασα 124. Με συγχωρείτε, εγώ φταίω να το ελέγξουμε. Νόμιζα ότι εγκρίθηκε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικώ. Πατήστε τα κουμπιά σα. 124. Πέρα. Σαφώ εγκρίνεται. 3 προ 31. Συμβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Επίσης εγκρίνεται. Τώρα 151. Εδώ έχουμε ένα σύνολο τροπολογιών. 151 έως 160. Ψηφίζουμε συνολικά. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτονται. Τώρα 39 40 και 41. Υπέρ. Κατά. Δεν είδα το ΕΛΚ. Ωραία. Ξανά, παρακαλώ. 39 έως 41. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 156 εκπαιδεύει, 42 και 43 μαζί. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνονται. 44 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 180 εκπίπτει. 184-185 υπέρ. Κατά. Απορρίπτονται. 186 πρόσθετη υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. Εγκρίνονται. 190 Άρχεται η ψηφοφορία. 190. Πέρας. Απορρίπτεται. 191. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 193. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 192 εκπίπτει. 194. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Άρθρο 46. 196. Υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 195. Υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 198. Υπέρ. Άρχεται η ψηφοφορία. 48 με συγχωρείτε, 48. 48 πέρας. Εγκρίνεται με 18-29. 50 τώρα. 50 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. ...201, 199 201, υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 202. Επέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Με διαφορά. 203 και 204. Υπέρ. Άρχεται η προφορία. για τις 203-4. Πέρας. Απορρίφθηκε με μία ψηφοδιαφορά. 205. κυρία Ρούλε Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Κάνατε λάθος. άρχιτε τη ψηφοφορία για την 205. Πέρας. Εγκρίθηκε με μια ψηφοδιαφορά. 51. Εκπίπτει. 206 υπέρ κατά Αποχέ. 52 υπέρ κατά εγκρίνεται. 53 υπέρ κατά εγκρίνεται. 54 υπέρ κατά εγκρίνεται. 55 υπέρ κατά εγκρίνεται. 207 του κ. Μάντερ υπέρ κατά απορρίπτεται. 209 υπέρ Κατά. Εγκρίνεται. Μερικές από αυτές εγκρίνονται αυτομάτως. από την 170 η 56 λοιπόν, πάμε στην 56, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 211 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Και μετά συνολική ψηφοφορία, 57, 58, 59 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τώρα πηγαίνουμε στην 17 της Επιτροπής Μεταφορών. Υπέρ. Νομίζω να κάνουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία. 17 Επιτροπής Μεταφορών, άρθρο 18. Πέρας. Απορρίπτεται. Παραρτήματα. 62 και 18 της Επιτροπής Μεταφορών. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 221 υπέρ κατά απορρίπτεται. 230 υπέρ. Με συγχωρείτε, 220 υπέρ κατά εγκρίνεται. 66 υπέρ κατά εγκρίνεται. 71 υπέρ κατά εγκρίνεται. 72 υπέρ κατά Επίσης εγκρίνεται. Τώρα, σύνολα, 230, 34, 35, 36, 37. Υπέρ, κατά, απορρίπτονται. 232-238 του κ. Μάντερς, υπέρ. Επίσης απορρίπτονται. Τώρα πάλι σύνολο 241 έως 251 υπέρ, κατά, απορρίπτονται όλες. Κρίμα. 242 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 242. Να το ελέγξουμε. 242. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με μια ψηφοδιαφορά. φορά. 244. 244. Υπέρ. Άρχεται η ψηφοφορία μάλλον. Πέρας. απορρίπτεται διότι υπήρχε διαφορά στην ψηφοφορία. Πρέπει να επιταχύνουμε λίγο. Να πιέζετε μέχρι να ανάψει το κουμπί. Αυτή είναι η συμβουλή μου. Συμβαστική 6 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τώρα 280. Όχι, με συγχωρείτε, παράδειγμα 6, 80. Υπάρχει προφορική τροπολογία Ψηφίζουμε λοιπόν μαζί με την πληροφορική τροπολογία υπέρ, κατά, εγκρίνατε. Η ίδια τροπολογία χωρίς την προφορική αυτή. 271 της κυρία Ρουίλερ. 271 υπέρ. Νομίζω να ψηφίσουμε ηλεκτρονικώς για 271. Πέρας. Απορρίπτεται. 272 της κυρία Ζωήλα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με μία ψήφο διαφορά. 275 του κυρίου Σβάμπ υπέρ κατά Απορρίπτεται. 284 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 79 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά. απορρίπτεται. Ε, εγκρίνεται με διαφορά. Συμβαστική 8 με κατά τμήματα ψηφοφορίε. Περίπλοκο. Τέσσερα τμήματα. Συμβαστική του ΕΛΚ, Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και αυτή. Πρώτο τμήμα. Πρώτα. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τέταρτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Επίσης εγκρίνεται. Τώρα πάμε στην πρώτη τροπολογία. Πρώτη τροπολογία της αιτιολογικής σκέψης από τον εισηγητή. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τρία, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 96. Άρχεται η ψηφοφορία για την 96. Πέρας. Απορρίπτεται με μία ψήφο διαφορά. Να δούμε ως σύνολο τις τροπολογίες της Επιτροπής Μεταφορών. Κύριε Σιγητά, μπορούμε. 2, 3 και 4 λοιπόν συνολικά. Άρχεται η ψηφοφορία, νομίζω. Έναρξη της ψηφοφορίας για τις 2, 3, 4. Απορρίπτονται. 98 υπέρ κατά απορρίπτεται. 99 της κυρίας Ρουίλε υπέρ. Άρχεται μάλλον η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 4 του ιπέρ, υπέρ κατά εγκρίνεται. 6 του εισηγητή υπέρ κατά εγκρίνεται. 102 υπέρ κατά εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά εγκρίνεται. 5 ε, της Επιτροπής Μεταφορών υπέρ κατά εγκρίνεται. 9 υπέρ κατά εγκρίνεται. Και 105 υπέρ κατά Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα το σχέδιο έκθεση συνολικά. Άρχεται η ψηφοφορία για το σχέδιο έκθεση. Κάποιος έχει εισαγάγει την κάρτα του και δεν ψήφισε. Εντάξει. Πέρας. Εγκρίνεται με 28 υπέρ, 3 αποχές και καμία ψήφο κατά. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Φαντεκάμπ. Θα περιμένουμε τις περαιτέρω εξελίξεις για τη μελέτη δικτύπου και τα υπόλοιπα ζητήματα. Σας ευχαριστώ λοιπόν και τώρα περνάμε στην ψηφοφορία για τις επόμενες χρήσεις ορφανών έργων. Ο λόγος ε, στον Αντιπρόεδρο, στην Αντιπρόεδρο μάλλον, για το υπόλοιπο μέρος των ψηφοφοριών. Εγώ θα χρειαστεί. Να. Απουσιάσω λοιπόν επιτρεπόμενες χρήσεις ορφανών έργων. Είσαι και ο κύριος Μάντερς. έκθεση τη επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Κύριε Μάντερ, θέλετε να πείτε κάτι πριν την ψηφοφορία ή να αρχίσουμε. Να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για την αρμονική συνεργασία μας. Ωραία λοιπόν, ψηφίζουμε απευθεία. Η 54 της κυρίας Πρέντεγκας θα έχει αποσυρθεί. 8 του εισηγητού. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνατε. 55 ως προσθήκη του κ. Φόξ. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 56. Πέντεκαστ. Ως προσθήκη υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 57 της κ. Ρόδροπα. Υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 58 Σάλτεμοζε. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 9 του κύριο Μάντερ. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 59 εκπίπτει. 60 και 62 εκπίπτουν. Η 60 επίσης εκπίπτει νομίζω. Ωραία αποσύρθηκε. 63 τώρα. Το κύριο Ζουβάν και τη κυρία Γκαλό. Επέρ. Κατά. Απορρίπτονται. 64 και 65. Άρχεται η ψηφοφορία για τις 64-65. Πέρας. Εκρίνονται με 22 ψήφους υπέρ, τα κατά 10 ε, ε, με προφορική τροπολογία του εισηγητή σε δύο τμήματα. Όπως το λέει και ο κατάλογος προφοριών. Υπέρ για το πρώτο τμήμα. Κατά εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα τώρα. Άρχεται η ψηφοφορία για το δεύτερο τμήμα. Πέρας. Εγκρίνεται. 17 ψήφοι υπέρ, 13 κατά. 10 εκπίπτει. 66 εκπίπτει επίση. 67. Πρώτο τμήμα. Ψηφίζουμε μόνο για το πρώτο τμήμα. Συμβατώ με την τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά. Αγκρίνεται. 68. Υπέρ. Κατά. Αγκρίνεται. 69. Υπέρ. Κατά. Αγκρίνεται. Συμβαστική 1. Υπέρ κατά εγκρίνεται. 71 της κυρίας Σαλτεμόζε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται με διαφορά. 72 της κυρίας Σαλτεμόζε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω να ελέγξουμε ηλεκτρονικώς. 72 της κυρίας Σαλτεμόζε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται με διαφορά. 73 καλύφθηκε από τη συμβαστική, 74 της κυρίας Πέντεγκαστ. 74. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 12 με προφορική τροπολογία του κ. Μάντρης. Περ. Κατά. Αγκρίνεται. 75 και 77. Άρχεται η ψηφοφορία για τις 75-77. Πέρας. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται μάλλον. 76 της κυρίας Ρόιτοβα υπέρ κατά εγκρίνεται. 13, 13 αποσύρεται, 78 υπέρ κατά εγκρίνεται. 79 του κ. Φόξ υπέρ κατά εγκρίνεται. 80 81 υπέρ κατά εγκρίνεται. 82 υπέρ κατά εγκρίνεται. 83 υπέρ κατά επίσης εγκρίνεται. 84 και 85 μαζί. Άρχεται η ψηφοφορία για τους 84-85. 84, 85, 86 νομίζω μπορούμε να τις ψηφίσουμε συνολικά. Ναι, 84, 85, 86, 87. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Η 14 αποσύρεται. 88. 88. Άρχεται η ψηφοφορία για την 88. Πέρας. Απορρίπτεται και αυτή. 89. 89 υπέρ. Νομίζω πάλι πρέπει να ψηφίσουμε ηλεκτρονικός. 89. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Είναι 15 αποσύρεται, 90 επίσης, 91. Με προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Με διαφορά. Η 91 εκπίπτει, 92 του κ. Φόξ. Υπέρ. Να ψηφίσουμε. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 92. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται με διαφορά. Με 93 με προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η 94 γλωσσική. 95 του κυρίου Έκστρομ. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 96 της κυρίας Ζόιτοβα υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 97 του κυρίου Πάξα υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 98 της κυρίας Πέντεγκαστ, κατά, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Αιτιολογικές σκέψεις 16 καλύφθηκε, 17, 18, 19, υπέρ, κατά, εγκρίνονται. Και τώρα πάμε στην 23. Τροπολογία 23, γιατί άλλε καλύφθηκαν. 23 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 24 ως προστίκη. Η 23 εγκρίθηκε υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 25-26 αποσύρονται, 27 είναι γλωσσική, 28 υπέρ. Με την κυρία Γκαλό και τον κύριο Ζουβά. Άρχεται η ψηφοφορία για την 28 με την προφορική τροπολογία της. Πέρας. Απορρίπτεται. Πρέπει λοιπόν να ψηφίσουμε τυπικώς την 28 χωρίς την προφορική τροπολογία. Η 28 λοιπόν ψηφίζεται χωρίς την προφορική τροπολογία. Απορρίπτεται. Είναι σαφέ. Α το ελέγξουμε. 28 υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. Με 29 υπέρ, κατά. Εγκρίνεται. Πηγαίνουμε τώρα στην τροπολογία 2 του κ. Μάντερ. Υπέρ, κατά. Εγκρίνεται. 33 ως προστίκη. Εντάξει, αποσύρθηκε. και 3 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 37 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τώρα πηγαίνουμε στην 42 της κυρίας ΣΑΛΤΕ Μόζερ. Άρχεται η ψηφοφορία για τον 42. Πέρας. Απορρίπτεται. 48. με προφορική τροπολογία. 48 με προφορική τροπολογία υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 47 ως προσθήκη στην 48, υπέρ, κατά, Εγκρίνεται επίση. 46 ω προσθήκη επίση. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται και αυτή. Τροπολογία του κυρίου Γιόγκ, 49 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται με διαφορά. Δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία για το δεύτερο τμήμα. Πέρας. Απορρίπτεται. Μια μικρή διαφορά. Η συμβαστική 2 στην αιτιολογική σκέψη 20 κάλυψε τις τροπολογίες 50-51 και 6 πηγαίνουμε στην 52 τώρα του κυρίου Μάντερς. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 53 με προφορική τροπολογία της κυρίας Πέντεγκαστ. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Και 53 εκπίπτει. Ψηφίζουμε λοιπόν τώρα τελική ψηφοφορία για το σχέδιο έκθεση. Άρχεται η ψηφοφορία για το σχέδιο έκθεση. Πέρα. 30 ψήφοι υπέρ, καμία κατά. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Μάντερς. that finishes the voting? Yeah. Right. So that concludes the voting and I'm now going to hand over to Mrs. Εδώ ολοκληρώνεται η ψηφοφορία και θα παραδώσω την προεδρία στην κυρία Βερνιό. ¿Todo el mundo está sentado? <laughs> ¿Preparado? Όσοι είναι να φύγουν ναι, να το πράξουν σιγά σιγά. Συνεχίζουμε λοιπόν. Καλημέρα σε όλες και όλους. Περνάμε με την απαλλαγή του, του γενικού προπολογισμού, το τμήμα 3 του 2010. Είναι ο κύριος Μπουσόη αυτός ο οποίος είναι εισηγητής. Θα του δώσω το λόγο και θα μας δώσει ένα νέο χρονοδιάγραμμα. Αν κατάλαβα καλά, παρακαλώ έχετε μέσα το λόγο. Θα συνεχίσω στα αγγλικά. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα έγγραφα που μας έστειλαν, για την καλοσύνη που είχαν να απαντήσουν στις γραπτές μας ερωτήσεις, για να ελέγξουμε τους λογαριασμούς τους και να δώσουμε την απαλλαγή. Πρέπει να σας πω ότι είναι περίπλοκο το θέμα και η άσκηση αυτή, γιατί πρέπει να κοιτάξουμε πολλά πράγματα, αλλά και απολύτω απαραίτητη για να δούμε τι γίνεται με την εκτέλεση των προπολογισμού σε θέματα που μας αφορούν ε, προστασία των καταναλωτών και νέα αγορά και αν αυτό δεν ισχύει τι μπορεί να γίνει για να διορθωθεί. Είναι πολλά τα θετικά ως προς τη δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα που άπτονται του ενδιαφέροντος τη Επιτροπής μας. Καταρχάς θα πρέπει να αναγνωρίσουμε τη σημαντική βελτίωση που έχει σημειωθεί στο Europortal που είναι μια ενιαία θύρα πύλη εισόδου για να γνωρίζουν οι πολίτες τα δικαιώματά τους και οι επιχειρήσεις τα δικαιώματα που απορρέουν από την εσωτερική αγορά. Η Επιτροπή μας παγίως το ζητούσε αυτό και μπορώ να σας πω ότι χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έχει λάβει υπόψη της. Αντιστοίχως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε να ε, έχει ένα μηχανισμό τύπου Solvit και U-Pilot για την εναλλακτική επίλυση των διαφορών. Και εδώ έχει γίνει πρόοδος, αλλά θα καλούσα την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειες, γιατί έχουμε ακόμα πρόβλημα συνειδητοποίησης και ενημέρωση και των πολιτών και των επιχειρήσεων. Και αν θέλουν όλοι να απευθολούνται από την ενιαία αγορά χρειάζεται προσπάθεια. Σε ό,τι αφορά το δίκτυο ECC, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε μελέτη εντεκτύπου για να μετρηθεί η αποτελεσματικότητα. Το καλωσορίζουμε και αυτό. Έχουμε ήδη τα στοιχεία και τα αποτελέσματα της έρευνας. Χρειάζεται μελέτη τώρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λήψη μέτρων για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα του δικτύου και να χρηματοδοτείται σωστά. Και πάλι θα πρέπει να γίνουν περισσότερες προσπάθειες για να αυξηθεί η προβολή και η γνώση των πολιτών σε αυτά τα θέματα και το δίκτυο. Επιπλέον, χαίρομαι που αυξήθηκε η εκτέλεση των πιστώσεων πληρωμών σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Αν δούμε ως λογαριασμούς στη Γενική Διεύθυνση ε, Υγείας και Καταναλωτών, σε πολλούς τομείς έχει ε, αρμοδιότητες αυτή η Γενική Διεύθυνση, αλλά ο τομέας των καταναλωτών ε, ε, έχει τη μικρότερη απορρόφηση των πιστώσεων. Μας λένε ότι η δικαιολογία είναι ότι είχαν υπερεκτιμηθεί οι ανάγκες. Αν χρειάζεται αυτό να το εξετάσουμε και πάλι και να υπάρχουν πιο ρεαλιστικές εκτιμήσεις για τις πληρωμές στο μέλλον. Τέλος, χωρίς αυτό είναι λιγότερο σημαντικό, να πω δύο λόγια για την τελωνιακή πολιτική. Χαίρομαι για τον εξυγχρονισμό του τελωνιακού κώδικα και τον τρόπο με τον οποίο το εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παραδέχομαι ότι δεν είναι καθόλου εύκολο. Έχει καθυστερήσει λίγο, αλλά το, ξέραμε. Και πάντως χρειάζεται να έχουμε πιο ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα και ε, πραγματικά παροτρύνω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει υπόψη της ε, τις ειδικές συστάσεις ε, που κάνουμε για τα τελωνία στην έκθεση που μόλις ψηφίσαμε. Επίσης και το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο ε, δείχνει ε, στην έκθεσή του ότι υπάρχουν κάποιες παρατυπίες ε, στις δηλώσεις των κρατών μελών, κυρίως στο θέμα των ιδίων πόρων. Υπάρχει υποκαταβολή των ιδίων πόρων σε πολλές περιπτώσεις. Ελπίζουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πιέσει τα κράτη-μέλη ώστε να διορθωθούν αυτές οι καταστάσεις και να αποφευθούν στο μέλλον. Όπως ορίζει το ελεκτικό συνέδριο, καλό θα ήταν να αποφεύγονται σφάλματα σε ποσά των ε, παραδοσιακών ιδίων πόρων. Αυτό θα γίνει με ε, γερούς ε, και σωστούς τελωνιακούς ελέγχους για να συλλέγονται σωστά οι δίπολοι. Για το χρονοδιάγραμμα τώρα, θα ήθελα και αυτό να σας το παρουσιάσω, έχω την εξή πρόταση. Σχέδιο γνωμοδότησης θα φύγει αυτή την εβδομάδα για να πάει στη μετάφραση κυκλοφορεί στα αγγλικά και θα αποσταλεί και ε, στους ε, σχεδόν και όσους άλλους συναδέλφους ενδιαφέρονται. Προτείνω στις 24-25 Ιανουαρίου να συζητήσουμε το σχέδιο έκθεσης ανάλογα ε, με το τι θα αποφασίσει ο πρόεδρος ή η γραμματεία για να ψηφίσουμε στις 6 Φεβρουαρίου. Αυτά και σας ευχαριστώ πολύ και προσβλέπω στα σχόλια και τις προτάσεις των συναδέλφων. Ευχαριστώ πολύ. Επαληθεύσατε για την ψηφοφορία στην Επιτροπή 6 Φεβρουαρίου, αν δεν κάνω λάθος. Μήπως χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο. Δεν έχουμε, συνήθως δεν έχουμε πολλές τροπολογίες για την απαλλαγή μόνο. Αν επιμένετε όμως, θα μπορούσαμε να έχουμε μια έξτρα συνεδρίαση να συζητήσουμε τις τροπολογίες, να δούμε το σχέδιο γνωμοδότησης και μετά να ψηφίσουμε. Ο κύριος Ντάν τώρα ίσως να, να σας πει κάτι παραπάνω. Αλλά αυτά είναι που προτείνω εγώ, πρόεδρος. Όπως θα προτείνατε λοιπόν. Και θα δούμε αν στην πράξη υπάρξουν δυσκολίες τότε αν όπως πέρσι δεν πάρξουν τότε καλώς. Λοιπόν, το λόγο στους σκιώδεις εισηγητές Ο κύριος Σφάμπ απουσιάζει, αλλά θα πάρει το λόγο ο κύριος Άριας Τσεβερία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εξ του σχεδίου συζητητού του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο, του κύριου Σφάμπ, θέλω να σας πω μόνο ότι συμφωνούμε απολύτως σχεδόν ε, 100% με τις προτάσεις του συντάκτης γνωμοδότησης. Δεν έχουμε να προσθέσουμε τίποτα παραπάνω. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα. Υπάρχει τώρα αντιπρόσωπος της κυρίας Σαλντεμόζε on, me fait <laughs> you, θα ε, μιλήσω Εγώ είμαι σκιώδης ή συγγέτρια. Δεν είναι ο Κρίστερ. Θα, όπως και ο προηγούμενος ομιλητής, θα ήθελα να πω, δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι περαιτέρω. Θα περιμένουμε το σχέδιο γνωμοδότησης από, γνωμοδότηση από τον εισηγητή και μετά θα επανέλθουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την Άννα. Θα περιμένουμε λοιπόν. Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω να προσθέσουμε. Ε, ε, δεχόμαστε τις ε, θέσεις του εισηγητή. Για τους πράσινας τώρα κάποια σχόλια. Η κυρία Χάιντι Ρούλε. Ναι, το ίδιο ισχύει και για μένα. Με <laughs> όλους τους προλαλήσαντες. Καλές οι προτάσεις του κυρίου Μπουσόη και θα τον υποστηρίξουμε. Για την ΚΟΕ τώρα. Θα δώσω το λόγο για το EFD. Κύριο Σαμβινί, δεν τον βλέπω ούτε και αυτόν. κάποιο άλλο από την ομάδα του, όχι. Δευτέρα απόγευμα, τι να πω. Άλλοι που δεν είναι οι εισηγητές, μήπως θα επιθυμούσαν να, να πάρουν το λόγο, έχουν το δικαίωμα. Παρακαλώ. Κανείς. Και όμω είναι ένα σημαντικό θέμα το θέμα της απαλλαγή για το γενικό προπολογισμό. Θα δούμε τον Γενάρη λοιπόν. Αν κανείς δεν θέλει τώρα να σχολιάσει, έχοντας αποφασιστεί το χρονοδιαγράμμα από τον κύριο Μπισόη, περνάμε στο επόμενο μας θέμα, το οποίο και αυτό είναι του κυρίου Μπισόη. Παρακαλώ, έχετε ξανά το λόγο. Κρισιάν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας μιλήσω τώρα για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020, που είναι από τα σημαντικότερα θέματα που έχουμε φέτος να συζητήσουμε. Εγώ επικεντρώθηκα σε κάποια θέματα που έχουν να κάνει ακριβώς με θέματα της ε, δικής μας Επιτροπής εσωτερική αγορά και προστασία των καταναλωτών. Πιστεύω ότι το επόμενο πολιετές πλαίσιο θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για να φτάσουμε στους στόχους πολιτικής που έχουμε ήδη ορίσει ή θα ορίσουμε τους επόμενους μήνες. Είναι χρήσιμο επίσης για τους στόχους στρατηγικής ε, για το 2020 και την ανάκαμψη της οικονομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διάβασα την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με μεγάλο ενδιαφέρον και πρέπει να σας πω ότι είναι πολλές ενδιαφέρουσες ε, όσο και καλές προτάσεις που περιέχει και συνδέεται και με τη στρατηγική του 2020 για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλωστε έτσι θα πρέπει να είναι προτείνουν κάποιες διαρθρωτικές αλλαγές, κοινά στρατηγικά προγράμματα, το καλωσορίζω αυτό πάρα πολύ, ε, ποντάρει στην έρευνα και στην ανάπτυξη, στα διαρθρωτικά ταμεία, απλούστευση των διαδικασιών για τους δικαιούχους. Υποστηρίζω πάρα πολύ αυτή την προσπάθεια ολόψυχα και ελπίζω τα κράτη-μέλη που θα έχουν τον τελικό λόγο να δείξουν ευαισθησία και να μην μπουν στον πειρασμό να περικόψουν την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κατά την άποψή μου, αυτό το πολιετές πλαίσιο θα πρέπει να επικεντρωθεί σε τομείς πολιτικής, όπου υπάρχει πραγματική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και μπορεί πραγματικά να κάνει τη διαφορά η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σύγκριση με δράση μεμονωμένων κρατών μελών. Να σας δώσω μερικά παραδείγματα που θεωρώ πάρα πολύ σημαντικά και πάρα πολύ σύντομα. Το επόμενο λοιπόν πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο θα πρέπει να επικεντρωθεί στην έρευνα και την καινοτομία, που μπορεί να τονώσει σημαντικά σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία την ε, ανταγωνιστικότητά μας. 80 εκατομμύρια για το νέο ορίζοντα 2020 ε, είναι αύξηση 46% σε σχέση με το ισχύον πλαίσιο ε, και την περίοδο 2007-2013. Αυτό είναι πολύ καλό για την τόνωση της καινοτομίας όπως επανειλημμένως ζητούμε και στην πράξη για την ενιαία αγορά. Το πλαίσιο επίσης θα πρέπει να δώσει ένα μέσο στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που είναι πάρα πολύ σημαντικές για την ανάπτυξη της οικονομίας μας. Γι' αυτό επίσης θεωρώ πάρα πολύ χρήσιμο να δημιουργηθεί ένα ξεχωριστό πρόγραμμα που να έχει να κάνει με ε, την επαγγελματική ε, ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων και με βασικές δομές ε, που σημαντικά συμβάλλουν στην ανάπτυξη ενιαίας αγοράς. Και εδώ Μιλώ για υποδομές ενέργειας, μεταφορών ε, που ε, θα τονώσουν το εμπόριο σε υπηρεσίες και ε, αγαθά και στην ευρυζωνικότητα. Επίσης, στο μέσο η διευκόλυνση Connecting Europe, διασυνδέοντας την Ευρώπη. Πολύ θερμά υποστηρίζω την πρόταση αυτή της Επιτροπής. Προτείνει 40 δις για ε, τη δυνατότητα, αλλά οι ανάγκες είναι πολύ υψηλότερες. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι θα πρέπει εκτός από το προπολογισμό να βρούμε άλλα καινοτόμα μέσα χρηματοδότησης που να βασίζονται στη μόχλευση. Ε, ο Επίτροπος Νταλή επίσης ε, προτείνει ένα νέο πρόγραμμα προστασίας των καταναλωτών 2014-2020 που θα είναι πολύ σημαντικό για δράσεις που θα ε, δίνουν ε, περισσότερες δυνατότητες ε, στους καταναλωτές τέλος, ο εξυγχρονισμός των τελωνίων. Τα επόμενα αιτή θα πρέπει να γίνει πολλή δουλειά για να εφαρμοστεί ο εξυγχρονισμένος κώδικας τελωνιακός με μηχανοργάνωση, με υπολογιστές για να μπορούν καλύτερα να συναντούν μεταξύ τους στα τελωνία. Αυτές είναι οι σημαντικότερες περιοχές που χρειάζεται να εστιάσουμε τις προσοχής μας στους επόμενους μήνες. Βεβαίως υπάρχουν και άλλοι τομείς που δεν ανέφερα, αλλά δεν, ε, όπως ξέρετε συνεργάζομαι πάρα πολύ στενά με τους και και μπορούν να κάνουν τις τροπολογίες τους ανά πάσα στιγμή. Στόχος μου ανέκαθεν ήταν και παραμένει να προχωρήσω στη συνένεση στην Επιτροπή μας, να στείλουμε ισχυρό μήνυμα στην Επιτροπή Προπολογισμών και ελπίζουμε να έχουμε ένα τελικό αποτέλεσμα που να αντανακλά τις απόψεις μας. Χρονοδιάγραμμα επίσης να σας προτείνω. Θα στείλουμε το σχέδιο στη μετάφραση ε, περί τα μέσα Ιανουαρίου του 2012. Βεβαίως μόλις υπάρξει η αγγλική έκδοση θα τη διανύμουμε πριν τις μεταφράσεις προτείνω το σχέδιο της έκθεσης να το συζητήσουμε στις 6 Φεβρουαρίου του 12 και να ψηφίσουμε στις 20 Μάρτιου. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς, ευχαριστούμε. Θα δώσω το λόγο. Για το Λαϊκό Κόμμα, σιώδης ηγητής, έχει... Θέλετε να πάρετε το λόγο. Ο κύριος Άριας Ετσεβερία. Εξ ονόματο κύρια κυρίας Σαρτόρη. Ευχαριστώ. Ναι, γνωρίζουμε όλοι ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι βασικός πυλώνας της οικονομίας μας και αυτό το στοιχείο μα απασχολεί όλους και έχουμε την πρόθεση να το βελτιώσουμε και να ε, διευκολύνουμε τη ζωή τους. Πιστεύω ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε γοργούς ρυθμούς Συμφωνούμε με το χρονοδιάγραμμα που προτείνει ο συντάκτη και δεν έχω να προσθέσω πολλά περισσότερα. Ευχαριστώ πολύ. Για το SD, ο Αντώνιο δεν είναι εδώ. Βλέπω ότι δεν υπάρχει κανένα άλλο για την ομάδα. Ε, ίσως θα μπορούσα να πάρω εγώ το λόγο. Συγχαίρω τον κύριο Μπουσόη. Έχει δείξει τα σημαντικά θέματα σε αυτή την πρόταση. Έχουμε, έχουμε να κάνουμε το φάκελο με την νεωτερικότητα και την έρευνα. Έχουμε επιμείνει πάνω σε αυτό, στο θέμα της ανταγωνιστικότητας. Κάτι που πρέπει να προσέξει η γυραιά Ήπειρος και να οδηγηθεί στην ανάπτυξη. 46% παραπάνω σχέση με άλλα προγράμματα είναι κάτι το θετικό και όπως είπε ο κ. Αριάς, θα ήθελα να αναφερθώ σε μια προτεραιότητα που έχει να κάνει με την αγωνιστικότητα τη βιομηχανία, το βιομηχανικό χώρο, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είναι εδώ αυτό το οποίο θα πρέπει να προσέξουμε όσον αφορά την απασχόληση στις χώρες μας, ούτως ώστε να υπάρχει μια απασχόληση ισορροπημένη, που η οποία ανταποκρίνεται στις συνθήκες για την κοινωνική συνοχή, για τις μεγάλες υποδοχές μας αναφέρεται τον, τον αριθμό 40 δισεκατομμυρίων. Ωραία, καλά είναι τα ποσά, αλλά σε σχέση με τις ανάγκες που έχουμε, Τίποτα δεν είναι σε σχέση κυρίως με την Ευρώπη τη κρίση. Κάτι θα πρέπει να κάνουμε, να συζητήσουμε μήπως μπορούμε να πετύχουμε καλύτερου καλύτερους Και νομίζω ότι η Επιτροπή θα σας υποστηρίξει σίγουρα ότι θα πρέπει να βελτιωθεί ο προπολογισμό όσον αφορά τα τελωνία. Είδαμε τα προβλήματα που υπάρχουν με, την, με τα παραπημένα προϊόντα, υπάρχουν θέματα ασφάλειας, η προστασία του καταναλωτή. Σίγουρα πάνω σε αυτό το θέμα θα πρέπει να εμβαθύνουμε το προβληματισμό μας. Και για το ΕΣΕΡ δεν βλέπω κανένα. Για τους πράσινους σίγουρα είναι η Χάιντε. Οπ, φεύγει. Πάει και αυτή. Για την άλλη φορά λοιπόν. Και για την ΚΟΕ δεν έχουμε τίποτα. Κανείς. Κάποιος άλλος που θέλει να πάρει το λόγο σε... πέρα από τους σκιώδες συζήτητες. Σήμερα βλέπω ότι γρήγορα γρήγορα τα τελειώνουμε τα θέματα. Μα έδωσε το χρονοδιάγραμμα ο κύριο Μπουσόη που μα φαίνεται ικανοποιητικό. Αν κανεί δεν έχει κάποιε επιφυλάξει, παρατηρήσει να κάνει. Έφτασε η κυρία Γκριπ, θα μπορέσουμε να περάσουμε στο δικό τη θέμα. Και τη δίνω αμέσω το λόγο. Euh, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σήμερα έχουμε να κάνουμε με το θέμα το οποίο έχει να κάνει με την, ε, την εταιρική διακυβέρνηση. Υπήρξε μια πράσινη βίβλος για το θέμα αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τη στιγμή μάλιστα που περνάμε αυτή τη μεγάλη κρίση. Είναι πολύ κατάλληλο εμείς σαν Ευρωβουλευτές να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορεί να δούμε αυτό το θέμα της διακυβέρνησης των εταιρικών. Όλα αυτά να μπουν στην καρδιά του προβληματισμού μας για την πραγματική οικονομία. Οι εταιρείε θα πρέπει και για τους εργαζομένους τους και για τους μετόχους τους και για τους πελάτες τους θα πρέπει να δημιουργήσουν μια εμπιστοσύνη σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όλα αυτά φυσικά μέσα στο πλαίσιο της κοινή ενιαίας αγοράς. Έχει δεθεί μια πράξη από την Επιτροπή, δόθηκε έμφαση όσον αφορά το θέμα της εμπιστοσύνη και ότι θα πρέπει να το ξαναδούμε αυτό το θέμα της διακυβέρνηση των εταιριών. Σε σχέση με την πράσινη βίβλο λοιπόν της Επιτροπής, εμείς θα γνωμοδατήσουμε και θα απαντήσουμε επί Επίσης η Επιτροπή, εκτός από την πράσινη βίβλο, έχει εδώ και μερικές εβδομάδες εγκρίνει κάποιες προτάσεις τον Οκτώβριο που έχει να κάνει με τις ευθύνες των εταιριών. Η γνωμοδότηση που σας προτείνω θίγει κάποια θέματα. Το πρώτο έχει να κάνει και μου φαίνεται σημαντικό για μένα ότι η διακυβέρνηση των επιχειρήσεων πρέπει σίγουρα να συμβάλλει στην αηφόρο ανάπτυξη στην εσωτερική αγορά, την πραγματική οικονομία να υποστηρίξει, ανάπτυξη. Επίσης, να διασαφινιστούν στρατηγικές οι οποίες θα είναι μακροπρόθεσμες, όχι βραχυπρόθεσμες. διότι υπάρχουν απειλές, θα πρέπει να διονυσούν οι επιχειρήσεις, να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους, διότι δεν υπάρχουν επιπτώσεις κυρίως στους μικρομετόχους και βλέπουμε τα πράγματα τα οποία αντιμετωπίζουμε σήμερα όσον αφορά το θέμα που έχει να κάνει με τις βαρχιπρόθεσμε επενδύσεις και προοπτικές. Μακροπρόθεσμες λοιπόν επενδύσεις. Επίσης, ένα, υπάρχει, το θέμα του, των διοικητικών συμβουλίων, που να υπάρχει μια σύνθεση εκεί η οποία ε, την προτείνουμε εμείς, η οποία πρέπει να είναι πιο πολύμορφη, να λαμβάνει υπόψη την κοινωνική διάσταση, ούτως ώστε να υπάρξει ένα σωστός διάλογος για, τις προσανατολ... για τους στρατηγικούς προσανατολισμούς και να δοθεί έμφαση στους επαγγελματίες ε, στο θέμα του μάρκετινγκ των πωλήσεων, ούτως ώστε τα διοικητικά συμβούλια να μπορούν να έχουν ένα προγραμματισμό με μια σωστή στρατηγική όσον αφορά την επιχείρηση, σύμφωνα με τις ανάγκες, τις πραγματικές ανάγκες της ε, αγοράς και φυσικά των καταναλωτών. Ένα τρίτο θέμα που θα ήθελα να θίξω εγώ όσον αφορά τη διαχείριση των επιχειρήσεων να επιμείνουμε ότι τα θέματα των αμοιβών θα πρέπει να είναι υπεύθυνε. Φυσικά να σέβεται κανείς εδώ πέρα την αρχή που έχει να κάνει με την ισότητα και την ίση αντιμετώπιση φυσικά των δύο φύλων, ανδρών και γυναικών. Σε αυτά, και αυτά μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκή νομοθεσίας. Επίσης, να υπάρχει ενισχυμένη συμμετοχή των εργαζομένων ίσως μέσω μετοχικής ε, ε, συμμετοχής, να το δούμε αυτό, ούτω ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη, μεγαλύτερο κίνητρο για τους εργαζομένους. Σίγουρα υπάρχει και το θέμα της διαφάνειας και μια εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά τη φύση των πληροφοριών που κοινοποιούνται στους μετόχους, κάτι το οποίο θα ήταν προς ε, αυτά και περιμένω με ενδιαφέρον τη συμβολή των συναδέλφων σήμερα ίσως ή αργότερα. Δεν βλέπω και τόσο πολύ σήμερα το απόγευμα. Ίσως συμμετοχή μέσω τροπολογιών. Ε, ευχαριστώ πολύ. Alors, là, nous Έχουμε σκιώδη εισηγητή ο οποίο έχει φτάσει μονο Η Μπάρμπαρα μάλλον είναι για την S&D. Δεν ξέρω αν έχει προετοιμάσει κάτι. Αν θέλει, τη δίνω αμέσω το λόγο. Κυρία Βάιλερ από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, συγγνώμη που άργησα, αλλά έχω μια αντιπροσωπεία 35 Βιετναμέζων αυτό τον καιρό και καταλαβαίνετε. Ε, και είναι και στην άλλη άκρη του κτηρίου. Κοίταξα την πρόταση της συναδέλφου Λεγκρίπ. Σωστά το λέω. Και δεν έχω βρει τίποτα να επικρίνω. Αλλά τη βρίσκω και πάρα πολύ ήπια και μαλακή την πρόταση αυτή. Σοφτ. Τώρα γιατί γελάτε εκεί κύριε στη γραμματεία ή με διάτε, εν πάση περιπτώσει η πρώτη μου εντύπωση ήταν, μα γιατί υπάρχει κανένας λόγος, αν τα λέμε τόσο στρογγυλωμένα όλα αυτά, τόσο ε, ανώδυνα και τόσο ωραία. Έχουμε ξανακάνει τέτοια έκθεση, ξέρετε, και ήταν πολύ πιο οξία, πολύ πιο εχμηρή και πολύ πιο στεναρή για την καλή διακυβέρνηση μόνο στα οικονομικά, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ήταν ενδιαφέρον που τότε επί της ουσίας αρμόδια ήταν η Οικονομική Επιτροπή, ενώ τώρα είναι νομική, ούτε αυτό είναι πολύ λογικό. Αλλά όταν συζητούσαμε αυτά τα θέματα λοιπόν για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ε, η γνωμοδότηση για την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, ήμασταν πιο στεναροί, πιο θαραλέοι. Τώρα ε, έχουμε την ίδια έκθεση όχι μόνο για την οικονομία, για όλες τις εταιρείες που είναι εισηγμένες στα χρηματιστήρια όλες τις μεγαλύτερες εταιρείες και αυτά που ζητάμε νομίζω έτσι είναι λίγο light, ξέρω εγώ, δεν χρειάζεται, δεν τα φοβάται κανείς, δεν τρομάζουν κανέναν. Ε, ας βάλουμε και καμιά απέτηση, έτσι, κάτι πιο σκληρό που να έχει σχέση με την κρίση, με την απώλεια εμπιστοσύνη που ζούμε και οι εταιρείε και οι διευθυντές των εταιρείων ε, έχουν ε, πρόβλημα, δεν έχουν εμπιστοσύνη στους πολιτικούς και τούμπαλοι. Γιατί θα πρέπει και οι εταιρείε κάπου να βοηθούν για την κοινωνική συνοχή. Από ό,τι βλέπω, μόνο δύο μέρες προθεσμία έχουμε ακόμα, αλλά θα καθίσω να σκεφτώ λίγο πώς μπορούμε να το εμπλουτίσουμε το κείμενο, να το στείλουμε στη νομική επιτροπή. Και γιατί η νομική, δεν σας εκπλήσει αυτό να δώσουμε κάποιες ε, έτσι, προτάσεις για σκέψη και να βγει μια ουσιαστική έκθεση συνολικά ως πακέτο. Αυτά. Merci, Barbara. Ευχαριστούμε την Μπάρβαρα. Σημερώζουμε τις απόψεις του. Ο Σμιτ, έχουμε, αλήψει, λείπει πολλοί κόσμος και βλέπουμε ότι ίσως σε λίγο φτάσει και ο Λεσμίτ. Α, θέλει να προσθέσει κάτι η Μπάρμπαρα. Ήθελα να πω ότι συμμερίζομαι τις απόψεις σου. Θα πρέπει να είμαστε πιο δυναμικοί. Η κρίση είναι παρούσα. Θα πρέπει να είμαστε σαφέστατοι και ξεκάθαροι. Μπάρμπαρα. Ναι. Έχω και μια παράκριση. ξανά κυρία Βάιλερ θα το επαναφέρω αυτό το αίτημα της ποσόστοσης στα διοικητικά συμβούλια των εταιριών. Και καλό θα ήταν να το παλέψετε, να το προωθήσετε. Η προηγούμενη έκθεση ήταν προεξαμήνου. Παρακαλώ να το υπερψηφίσετε γιατί αυτό βοηθάει τις εξελίξεις στην Ευρώπη. Je vais redonner la parole au rapporteur. το λόγο στον εισηγητή. Στην στην κυρία, συγγνώμη, εισηγήτρια. Oui, euh, Ευχαριστώ. Κάποιες... Ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις που γίνανε. Απλώς να πω ότι το τι σχέδιο, σε σχέδιο βρισκόμαστε ακόμα για τις συζήτησεις, θα έχουμε τις δυνατότητες, θα μπορέσω να συνεργαστώ και μετά τα Χριστούγεννα με τους σκιώδεις συζητές της το το σχέδιο είναι μια βάση για συζήτηση, για προβληματισμό. Η γνωμοδότηση λοιπόν που σας προτείνω σαν βάση ε, στηρίζεται σε έξι προτάσεις. Για το, τη σύνδεση των συμβουλίων διοικήσεις, για τα θέματα των, των, της ισότητας όσον αφορά τις αμοιβέ, για τους εργαζόμενους, για την ενημέρωση που γίνεται προς τους μετόχους, η οποία θα μπορούσε να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συγκεκριμένες προτάσεις κάνω, αλλά σίγουρα πήρα το μήνυμα που μου δόθηκε. Θα σκύψω πάνω από το ένα αβ θέμα, να είμαι πιο συγκεκριμένη και φυσικά να ήθελα να πω με πολύ ενδιαφέρον περιμένω τη συμβολή σας διότι είναι σαφέστατα όταν δουλεύουμε εδώ σε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσπαθούμε να προχωρήσουμε και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι πάντοτε μια σύνθεση. Ε, φυσικά καταλήγοντας σε ρεαλιστικές προτάσεις από τη μεριά των συναδέλφων. Βλέπω ότι ξαναμουζήτησε το λόγο η, κυρία, η Μπάρμπαρα. Ναι. Η κυρία Βάιλερ. Με το χρονοδιάγραμμα έχω μια παράκληση και πάλι. Με εκπλήσει πάρα πολύ που απουσιάζουν τόσο πολλοί σκιώδεις σήμερα και άλλοι ε, μέλη της Επιτροπής μας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Την εβδομάδα πριν τα Χριστούγεννα, βεβαίως δεν είχε προβλεφθεί συνεδρία Επιτροπής. Και τελικά διοργανώθηκε εκ των υστέρων. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να έρθω τότε. Δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα. Την άλλη εβδομάδα θα μπορούσα να βρω μία ωρίτσα ή μισή ώρα τουλάχιστον και πάνω. Αλλά παραμονές Χριστουγέννων δεν μπορώ να ξανάρθω στις Βρυξέλλες. Αναρωτιέμαι για την προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών Σήμερα είδαμε το, την πρόταση 8 Δεκεμβρίου, την Πέμπτη, είναι δυνατόν να είναι αυτή η προθεσμία. Δεν είναι καλό για, για τις εργασίες μας αυτό. Είχα προτείνει να προσθέσουμε άλλη μια εβδομάδα. Στο Στρασβούργο θα είμαστε Άρα μέχρι τότε οι σκιώδεις θα μπορέσουν να βρεθούν με την κυρία Γκριπ. Ε, αλλιώς την πέμπτη είναι πολύ μικρή. Συμφωνούμε? Καλώς. Okay. Προσέτουμε λοιπόν μια εβδομάδα. Παράταση. Οκτώ συν 7. Άρα 15. 14 τέλο πάντων. Κυρία Λεγκρίπ, θέλετε ξανά το λόγο. Σύντομα, για το χρονοδιάγραμμα. Η παράταση, μια χαρά, σωστή πρόταση, μου προτάθηκε από την Επιτροπή μας και νομίζω ότι όντως πρέπει να περιμένουμε ούτως ώστε κάποιοι συνάδελφοι που τους ενδιαφέρει αυτό το θέμα να το μελετήσουν, να δουν την γνωμοδότηση, να προσθέσουν ίσως κάποιες απολογίες. είχα προβλέψει μια, ε, πριν να τα μια συνεδρίαση, ίσως 20 Δεκεμβρίου, αλλά με βάση αυτό ήθελα να δω μήπως μπορούμε σαν να συναντηθούμε με τους οι εισηγητές. Αν υπάρχουν όμως δυσκολίες, μίζωνα σημασία, τότε καταλαβαίνω να προτείνουμε κάτι άλλο. Αλλά η Επιτροπή για, που είναι επί της νομικών θεμάτων 4, 4 Ιανουαρίου θα συναντηθεί. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτό το θέμα με την πρόταση της Πράσινης Βιβλίου της Επιτροπής θα πρέπει να ψηφίσει για τη συνολομέλεια το Φλεβάρι λοιπόν. Πρέπει να το λάβουμε υπόψη και αυτό. Ευχαριστώ. Λοιπόν, χρονοδιάγραμμα. Παράταση για τις τροπολογίες. Η Επιτροπή 20 Δεκεμβρίου θα συναντηθεί, η και θα ασχοληθεί με την απολογισμό της ε, Πολωνικής Προεδρίας. Λοιπόν, για τις 15 Δεκεμβρίου προθεσμία της απολογίας. Πώς μπορεί να ψηφίσει κανείς 9 Γενάρη την ΙΜΚΟ τη στιγμή που οι τροπολογίες έχουν προταθεί μόλις πριν από τις διακοπές. Άρα πρέπει να, και σε αυτό το θέμα να δώσουμε μια παράτηση. Η ψηφοφορία στην ΙΜΚΟ θα δούμε και από την Επιτροπή για τα νομικά θέματα μήπως και αυτοί μπορούν να δω, κάνουν μια παράταση. Είναι ένα σημαντικό θέμα. και με αυτόν τον τρόπο ίσως να μην ψηφίσουμε στην Ολομέλεια το Φεβρουάριο. Βλέπω όμως και τον κύριο Σμιτ που έχει καταφθάσει. Του δίνουμε το λόγο. Είναι η ητής για την φιλελεύθερους. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είστε ταχύτατε σε αυτή την Επιτροπή σήμερα. Υπήρξε ακρόαση στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, δεν ήμασταν τόσο γρήγοροι. Είμαι σκεώδης εδώ για την εταιρική διακυβέρνηση. Για αυτό το θέμα να μιλήσω ή το ολοκληρώσετε. Πολύ ωραία. Θα προσπαθήσω να υποθέσω ότι υπόθηκε και να κάνω κάποια σύντομα σχόλια. Ή το ενωσιακό πλαίσιο εταιρική διακυβέρνηση και ο κώδικα για την καλή διακυβέρνηση είναι πολύ σημαντικό εργαλείο, κατά την άποψή μου. Θα εξυπηρετήσει τις εταιρείε ώστε να ενισχύονται και να γίνονται ευφιέστερε. Και θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη στην ενιαία αγορά. Αυτό το χρειαζόμαστε, πιστεύω, στην Ευρώπη. Ιδιαίτερο στη σημερινή περίοδο. Βεβαίω, πρέπει να πετύχουμε μια ευαίσθητη ισορροπία μεταξύ ενό σαφού πλαισίου για την εταιρική διακυβέρνηση και την ποιότητά του και βεβαίω να επιτρέπουμε και στου κατόχου των εταιριών να λαμβάνουν τι δικέ του αποφάσει. Αυτό ανέκαθεν ήταν και θα συνεχίσει να είναι μια ισορροπία αρκετά δύσκολο να εξευρεθεί. Ω τώρα, πιστεύουμε ότι η αυτορύθμιση μπορεί να λύσει τα προβλήματα. Εγώ είμαι υπέρ αυτή τη λύση ε, σε γενικέ γραμμέ μεν, αλλά βλέπουμε ότι ίσως χρειάζεται να έχουμε αυστηρότερο πλαίσιο κανόνων. Ακόμη και έτσι όμως, ένα τέτοιο αυστηρότερο πλαίσιο θα πρέπει να είναι προσεκτικά σχεδιασμένο. Εδώ άκουσα την συγκεκριμένη αναφέρει την εκπροσώπηση των γυναικών. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Οι γυναίκες ανέκαθεν υπήρξαν μειονότητα και Πολύ συχνά μάλιστα στις πολιτικές ομάδες όπου εγώ υπηρέτησα. Ε, πιστεύω λοιπόν ότι είναι ουσιαστική σημασία να έχουμε αυστηρή ισορροπία μεταξύ των δύο φύλων και στις εταιρείε, σε όλες τις εταιρείε, όχι μόνον. Συνάδελφοι, γνωρίζετε, δεν είμαστε και τόσο πολλοί, τέλος πάντων γνωρίζετε ότι δεν υπάρχει καμία γυναίκα στο, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Γερμανίδα, όχι. Στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ίσως το πλέον σημαντικό θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα, μόνον άνδρες. Δεν έχω τίποτα κατά του κύριου Ντράγκη βεβαίω, αλλά θα, είχε, θα ήταν καλό να έχει μια γυναίκα στο πλευρό του. Αυτό ισχύει και για τις εταιρείε. Πρέπει λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί πώς θα σχεδιάσουμε αυτά τα μέτρα. Θα εξετάσω λοιπόν με πολύ θετική στάση τις προτάσεις σας για να δούμε πώς μπορεί να εξευρεθεί μια λύση σχετικά. Πάντως είμαι υπέρ των κανόνων, κανόνων που να μπορούν να εφαρμοστούν και σε δύσκολους καιρούς, όπως και σε πιο ηλιόλους τους για Ευχαριστούμε τον κύριο Σμιντ για τα σχόλιά του. Σαν γυναίκα συμμεριζόμαστε αυτά που είπατε. Παρόλο που δεν είναι δική μας αρμοδιότητα, δεν υπάρχει γυναίκα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πολλές φορές οι γυναίκες προτείνουν πολύ συγκεκριμένες λύσεις. Και θα ήταν καλό να υπήρχαν κάποιε γύρω από τον κύριο Ντράγκη. Κυρία Λεγκρή πάλι το λόγο, αν θέλει να κάνει κάποιο τελευταίο σχόλιο. Συμφωνώ και εγώ με τον συνάδελφο Σμιτ. Τον ευχαριστώ που έκανε θετικές, ε, ε, θετικά σχόλια σε σχέση με τα θέματα που βρουν την ισότητα όσον αφορά τα θέματα των δύο φίλων σε σχέση με τη μισολογία και φυσικά τη θέση γυναικών στα διοικητικά συμβούλια. Να συνεχίσουμε λοιπόν προς αυτή την κατεύθυνση, ξέροντας ότι ο, τρόπος με τον οποίο εκφράζει κανείς αυτές τις αρχές θα πρέπει να γίνεται με έναν τρόπο ρεαλιστικό και να κερδίσει την ευρεία υποστήριξη των ομάδων. Ευχαριστώ, Πρόεδρος. Είδαμε το χρονοδιάγραμμα και λέμε τροπολογίες 14 Δεκεμβρίου Τετάρτη. Κατάσταση τροπολογιών. Ουδέν σχόλιων από ό,τι βλέπω. Και περνάμε στον κύριο Σμιτ. Περνάμε κύριο Σμιτ στη δική σας την ε, εξέταση γνωμοδότησης. Σας δίνω αμέσως το λόγο Γρήγορα προχωρήσαμε κύριε Σμιτ, είναι αλήθεια. Α. Αλλά δεν είχαμε ε, έτσι μεγάλη διάρκεια διαλόγου διότι δεν είχαμε μεγάλη συμμετοχή. Παρακαλώ, τελευταίο θέμα έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εδώ έχουμε ενδεχομένως ένα από τα πλέον περίπλοκα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. όπως το ονόμαζα εγώ, ΚΕΘΔΕ, Κοινή Ενοποιημένη Φορολογική Βάση για τις εταιρείε. Γνωρίζουμε όλοι ότι η ιστορία αυτή έχει παρελθόν. Δεν επιλήθηκε επί σειρά ετών. Λίγο δύσκολο και τώρα να βρούμε λύσεις. Πάντως θεωρώ και θέλω να το τονίσω μιας αν και θα ήθελε να υπάρχουν εδώ εκπρόσωποι της Επιτροπής, έχει προσπαθήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βρει μια σωστή ισορροπία μεταξύ των αναγκών και του τι πρακτικά και πολιτικά θα έχει νόημα να προταθεί. Είναι εξαιρετικά ευαίσθητο ζήτημα. Οι ευρωπαϊκές ε, χώρες έχουν διαφορετικές φορολογικές βάσεις που λειτουργούν ως εμπορική φραγμή για την ανάπτυξη και την απασχόληση πρόταση για κοινή ενωπημένη φορολογική βάση θα οδηγήσει σε σημαντικέ ε, αλλαγέ στην φορολογική των εταιριών στην Ευρώπη. Με τη δυνατότητα να υπάρξουν βελτιώσει για τι εταιρείε που λειτουργούν διασυνοριακά, μειώνοντα το ε, φορολογικό βάρο και του ε, φραγμού που αυτή τη στιγμή επιβάλλονται. Καθώ και το κόστο. Όπω είπε και ο Επίτροπο, έτσι θα έχουμε μια αγορά πιο ενιαία και θα ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών εταιριών καθώ και την ελκυστικότητά του στο διεθνέ προσκήνιο. Συμφωνώ με αυτά. Όμω οι βασικέ μου ανασυχίες είναι ότι η κοινή ενοποιημένη φορολογική βάση θα πρέπει να είναι εθελοντικού χαρακτήρα για τι εταιρείε. Μπορεί κανεί να ονειρεύεται ένα δεσμευτικό υποχρεωτικό σύστημα, αλλά δεν νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα ήταν, πρέπει να είναι προτεραιότητα σήμερα. Ένα υποχρεωτικό σύστημα θα αυξήσει και το κόστο για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, οπότε δεν θα επιτρέψει την ανάπτυξή του και την ανταγωνιστικότητά του στην ευρωπαϊκή αγορά. Υπάρχουν εδώ λοιπόν ενέχονται κίνδυνοι. Επίσης, ε, θα πρέπει να σκεφτούμε και την ανταγωνιστικότητα την θεσμική. Δεν συνίσταται το σύστημα αυτό να γίνει υποχρεωτικό πριν να αποκομίσουμε πρακτική εμπειρία για το ποιε είναι οι συνέπειε τη λειτουργία του συστήματο. Επίση, το επίπεδο τη φορολογία θα πρέπει να είναι κάτι που θα αποφασίζεται από τα εθνικά κοινοβούλια. Αυτό είναι άκρα ε, σημασία. Στόχο εδώ είναι να ενισχύσουμε το σύστημα φορολόγηση των εταιριών, όχι όμω ε, να εναρμονίσουμε του φορολογικού δείκτε. Μιλάμε για μια πρόταση κοινή όλων στην συζήτηση. Μια παρατήρηση που για όλους ε, ο εναρμονισμένος φορολογικός δείκτης είναι μια ανησυχία που έχει λάβει υπέρματρες διαστάσεις. Επίσης θα πρέπει να αποφύγουμε τις απώλειες ε, εξ αρχής ώστε να ενισχύσουμε τις συνοριακές συναλλαγές των εταιριών. Η ε, ενοποιημένη αυτή φορολογική βάση θα πρέπει να ενισχυθεί και από την απλούστευση και να υπάρξει μια ενιαία θηρίδα για την εξέταση των σχετικών θεμάτων, ώστε να μειωθεί το γραφειοκρατικό άκθος και η φραγμή για το όλο σύστημα. Και για να μειωθεί το κόστος της συμμόρφωσης και για να υπάρχει μια κοινή ισότιμη μεταχείριση. Το σχετικό σύστημα θα πρέπει να είναι τόσο ελκυστικό, ώστε οι εταιρείε να επιλέγουν να συμμετάσχουν και να προκύπτουν από αυτό πραγματικά πλεονεκτήματα. Προτείνω, Πρόεδρε, τις εξής αλλαγές. Αλλαγές στην ε, φόρμουλα που προτείνεται, αυτή ίσως είναι και η πιο δραστική πρόταση, ο παράγοντα των πωλήσεων να μην χρησιμοποιείται αλλά η ενοποιημένη και κοινή φορολογική βάση να βασίζεται στην απασχόληση και τα περιουσιακά στοιχεία, το, δυναμικό, το ενεργητικό δηλαδή των εταιριών. Έπειτα, εφόσον ο προορισμό επιβάλλει μετατόπιση από την σημερινή αρχή τη απόδοση των φορολογικών δικτών στην χώρα πηγή, θα πρέπει εδώ να σκεφτούμε πώς ο φορολογικός δείκτη μπορεί να χρησιμοποιηθεί θεωρητικά από τι ευρωπαϊκέ χώρε και πώ τον αξιοποίησε και ο Σάς στην εκτόρα εργασία του. Επίση για τι μικρομεσαίε ε, εταιρείε που θα χάσουν φορολογικά, ε, ε, που δεν θα εμπίπτουν μάλλον σε αυτό το σύστημα, θα χαθούν και από σημαντικά φορολογικά εισοδήματα για τι διάφορε χώρε. Ευχαρίστω να ακούσω και τα σχόλια των συναδέλφων και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίση, Πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα φόρουμ για την ε, ενοποιημένη φορολογική βάση για τα κάτι μέλη ώστε να προελευθεί ένα σύστημα επίλυσης των διαφορών βάσει των άρθρων 126 και 123. Θα πρέπει μετά από τρία χρόνια να αναθεωρήσει την πρότασή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να δει ποιες είναι οι επιπτώσεις του άρθρου 133 της ΚΕΦΔΕ. Επίσης, θα πρέπει μετά από τρία χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δει ποια είναι τα υπέρ και κατά τη εισαγωγή ενό ενδεχόμενου υπερχρωτικού συστήματο και του να υπάρχει μια κοινή ενωπημένη φορολογική βάση για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πρόεδρε, στην πρότασή τη αναλύει και τι ενδεχόμενε συνέπειε τη οδηγία για τι φορολογικέ βάσει των 100 μελών, το εθνικό του εισόδημα και σε τοπικό επίπεδο. Συμπεριλαμβάνοντα κοινωνικέ και οικονομικέ διαστάσει ε, λόγω τη μετακίνηση οικονομικών δραστηριοτήτων και θέσεων εργασία εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η επέκταση τη πρόταση αυτή μπορεί να δημιουργήσει περισσότερε δυνατότητε συνεργασία και εταιρικών σχέσεων. Αυτέ είναι οι βασικέ αλλαγέ που προτείνω Ευχαριστώ να ακούσω τις παρατηρήσεις ε, των συναδέλφων. Αν όλα πάνε καλά, θα έχουμε ευρεία συνένεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σμιτ. Λοιπόν, κανονικά σκιώδες συγκητές με τη σειρά Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, κυρία Ρόιτοβα, θα καταφτάσει. Προηγουμένως εδώ ήτανε. Ξέρω ότι για σοσιαλιστές και δημοκράτες ο κύριος Λιμιόγνο θα έρθει στη συνέχεια. Θα δώσω το λόγο στο μόνο παρόντα, τον κύριο Ντε Είναι ένα θέμα το οποίο θα συζητήσουμε και με τους υπολείπους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα. Έχετε αμέσως το λόγο κύριε Ντουγιόγκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όντως, είναι πάρα πολύ δύσκολο το θέμα αυτό. Και ε, είναι τελείως διαφορετική η βάση ορισμένων ε, και άλλα λέει, ας πούμε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή Οσηγητής ή άλλα λένε μη κυβερνητικές οργανώσεις. Εγώ είμαι υπέρ μιας κοινής ενοποιημένης φορολογικής ε, βάση για να μην έχουμε αυτό που συμβαίνει σήμερα. Ορισμένες χώρες ε, έχουν προβλήματα που είχαν ε, πολύ ανταγωνιστική θέση και πλεονεκτήματα για τις επιχειρήσεις και έχουν τελικά φτάσει σε μια κατάσταση πολύ άσχημη και έχουν φτάσει περίπου και σε μηδενικό συντελεστή. Αυτό δεν είναι καλό. Αυτή τη φορά η πρόταση δεν είχε την πρόθεση να επιβληθεί ένας ελάχιστος φορολογικός συνελεστής σε όλη την Ένωση. Δεν είναι αυτό που συζητούμε. Δεύτερο μεγάλο πρόβλημα που έχουμε την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι και κάτι που θέλει ο συγητής ευχαρίστως, να παραμείνουν όλα αυτά σε εθελοντική βάση, δηλαδή να έχει μια επιχείρηση ποιο σύστημα θα υιοθετήσει. Ναι, αλλά αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα για τις εφορίες. Τα εθνικά φορολογικά συστήματα, πώς θα γίνει αυτό, θα γίνει ένα ευρωπαϊκό σύστημα και πώς θα προσαρμόζονται. Χρειάζονται και πόρους εκεί, ε, φοριακοί και προσωπικό και για την ίδια μου τη χώρα, την Ολλανδία, θα έχει τεράστιες συνέπειες. Διότι αν επιλέξουν επιχειρήσεις αυτό το σύστημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τότε εμείς θα χάσουμε 1,67% του ΕΠ μας. Είναι πάρα πολλά λεφτά αυτά, είναι τεράστιο ποσοστό, λόγω της ε, προσέγγισης που έχει επιλέξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επαναλαμβάνω, εγώ δεν θα είχα πρόβλημα με ένα ελάχιστο, με ένα χαμηλό κοινό συντελεστή, ε, αλλά ε, η Κομισιόν έχει διαλέξει άλλο δρόμο. Και αυτό τι σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις θα πληρώνουν λιγότερους φόρους, θα, επιλέγουν πού μπορούν να πληρώσουν λιγότερους φόρους. Δεν είναι καλό αυτό. Θα έρθουμε πολλές τροπολογίες, πάρα πολλές τροπολογίες, θα το δούμε πάρα πολύ σοβαρά το θέμα. Δεν ξέρω αν θα εγκριθούν όλες. Πάντως θα είμαστε πάρα πολύ σχολαστικοί και μεθοδικοί και οι τροπολογίες μας ε, θα έχουν στόχο να αποδομήσουν ή μάλλον να αλλάξουν τελείως την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οπότε μας περιμένει πάρα πολύ δουλειά και δύσκολη. Μάλιστα, ο Πρόεδρος. Και πολλή συζήτηση, όχι μόνο πολλή δουλειά. Θα δώσω τώρα το λόγο στο σκιώδιο εισηγητή των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, τον Λίμαν Γιώκ. Ευχαριστώ, Μπαναντέτ. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχω πάρα πολύ ανάμεικτα συναισθήματα σε αυτό το θέμα. Ω σοσιαλιστής και φεντεραλιστής ανέκαθεν ήμουν υπέρ της περαιτέρω μεγαλύτερης φορολογικής εναρμόνησης στην Ευρώπη. Οπότε καταρχήν συμφωνώ με μια κοινή ενοποιημένη φορολογική βάση ως ένα βήμα προς την εναρμόνιση του φόρου επιχειρήσεων. Πλην όμως, όταν διαβάζει κανείς την πρόταση οδηγία, διαπιστώνει ότι αυτό δεν είναι καθόλου στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το μόνο σαφές κίνητρο που προβάλλουν είναι να διευκολύνουν τη ζωή των επιχειρήσεων και των εταιριών που είναι παρούσες σε περισσότερα από ένα κράτη-μέλη και να κάνουν και οικονομίες οι εταιρείες. Λοιπόν, μεροληπτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει ποντάρει σε αυτό. Αφήνει σε κάθε εταιρεία τη διακριτική ευχαίρεια να επιλέγει αυτό το σύστημα ή όχι. Ή ε, το πιο συμφέρον σύστημα όπως είπε ο Ολλανδός συνάδελφος από την άλλη δεν λέει τίποτα το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ισορροπία που πρέπει να βρούμε ανάμεσα στη φορολόγηση της εργασίας και τη φορολόγηση κεφαλαίου ή πώς θα ελέγχονται καλύτερα φορολογικά οι επιχειρήσεις. Και κάτι που είναι πιο σοβαρό ακόμα δεν λέει τίποτα για την ανάγκη να καταπολεμηθεί το φορολογικό dumping ή τη φορολογική ε, μειοδοσία των κρατών μελών ε, σε ό,τι αφορά τη φορολόγηση των επιχειρήσεων το αντίθετο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, πρεσβεύει και υιοθετεί την ε, ε, ελεύθερη φορολόγηση των επιχειρήσεων και λέγει μάλιστα ότι είναι δύσκολο να προβλεφθεί η επίπτωση που θα έχει αυτό στα φορολογικά έσοδα των κρατών μελών και θα εξαρτηθεί τελικά από τους στρατηγικούς στόχους και επιλογές του κάθε κράτους. Δηλαδή, να κανονίσουν την πορεία τους στα κράτη-μέλη για να μην μειωθούν τα φορολογικά τους έσοδα. Να τα βγάλουν πέρα μόνα τους. Αυτό δεν στέκει ούτε πολιτικά ούτε οικονομικά. Είναι μεγάλες ανασφάλειες ως προς τα φορολογικά έσοδα και έρχεται εδώ να προστεθεί και το κόστος διαχείρισης ενός 28ου ε, εθελοντικού συστήματος φορολόγησης των εταιριών. Όταν ε, είναι αυτό προαιρετικό και χωρίς ένα ελάχιστο φορολογικό ε, συντελεστή σημαίνει ότι παίζουμε τους μαθητευόμενους μάγους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αγωνίζεται τώρα για να βγει από την πιο σκληρή και βαριά οικονομική κρίση όλων των εποχών. Ε, τα κράτη παλεύουν με ελλείμματα και με χρέη. Ορισμένοι θέλουν να ενισχύσουν το σύμφωνο σταθερότητας για να ελέγχουν τους κρατικούς προϋπολογισμούς και να τιμωρούν τους παραβάτες που δεν μπαίνουν σε αυτή την άσκηση ε, τη ε, δημοσιονομική και εμείς ε, ως βουλευτές ερχόμαστε λέει να ψηφίσουμε για θέματα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ομολογεί ότι δεν έχει ιδέα για το τι επιπτώσεις θα έχουν αυτά στα οικονομικά και στα έσοδα των κρατών μελών. Δίνει λοιπόν προτεραιότητα σαφέστατα στα συμφέροντα των επιχειρήσεων Ευρωπαϊκή Επιτροπή εις βάρος των δημοσίων οικονομικών και της κοινωνικής δικαιοσύνης και της φορολογικής και εις βάρος των πολιτών που πλήττονται σκληρά από τη σημερινή κρίση. Ο μόνος τρόπος η κοινή ενωπημένη φορολογική βάση να είναι πρόοδος θα, θα ήταν να υπάρχει ένας ελάχιστος φορολογικός συνελεστής, να είναι υποχρεωτική και όχι αναδρομική ισχύς. Θα μπορούσαμε να εμπνευστούμε ε, από το σύστημα ε, το νομισματικό, το ΦΥΔΙ θυμάστε το 1972, και να διανέμονται τα κέρδη και τα ωφέλη μεταξύ των κρατών μελών. Στο σχέδιο έκθεσης ε, ο εισηγητής δεν αμφισβητεί ε, ούτε τον εθελοντικό χαρακτήρα του συστήματος, ούτε την έλλειψη ελάχιστη του φορολογικού συντελεστή και έχω απογοητευτεί γιατί νομίζω ότι ορισμένα από τα θέματα αυτά τα εστερνιζόταν. Κάνει λόγο για μια φόρμουλα μαθηματικό τύπο διανομής των εισόδων, κωδικοποίησης. Εντάξει, αυτό το καταλαβαίνω, αλλά ομολογώ ότι πολύ δύσκολα θα βρούμε τη σωστή φόρμουλα γιατί θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό αυτό από τον τρόπο με τον οποίο θα αντιδράσουν ε, οι εταιρείε. Αυτή όμως είναι μία παράμετρος μεταβλητή την οποία αγνοούμε. Επίσης γίνεται λόγος για αναθεώρηση ε, τρία έτη παρακαλώ, με μια τριετία μετά από την θέση ισχύ και όχι πενταετία όπως προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ Λίμ, λέει Πρόεδρος, για αυτή την πλήρη περιγραφή και ανάλυση της κατάστασης. Θα επανέλθουμε στο χρονοδιάγραμμα γιατί και εδώ, όπως και στο προηγούμενο θέμα και πολύ περισσότερο, γιατί γίνεται συζήτηση και υπάρχει ανάγκη συζήτηση στις ομάδες, θα χρειαστεί να αλλάξουμε το χρονοδιάγραμμα. Η κυρία Ρόιτο και ο από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Δυστυχώ επειδή άλλαξε το ωράριο συζήτηση, δεν ήμουν εδώ από την αρχή, δεν άκουσα τον εισηγητή και του Κιώδη, γιατί βρισκόμουν σε άλλη συνεδρίαση. Όμω, σε γενικέ γραμμέ, πρέπει να πω ότι είμαι υπέρ τη ε, πρόβλεψη μια ενοποιημένη φορολογική βάση, κυρίω για να εξυπηρετήσουμε του επιχειρηματίε, τι εταιρείε και να πατάξουμε τη φοροδιαφυγή. Καλό θα ήταν να ενοποιηθούν και να εναρμονιστούν οι φορολογικές εκτόσεις, να ευθυγραμμιστούν οι φορολογικές διατάξεις και να προσπαθήσουμε να επιτελέσουμε πρόοδο. Εδώ ε, συμφωνώ με τον εισηγητή ότι θα πρέπει να είναι τουλάχιστον προαιρετική συμμετοχή σε αυτό το σύστημα για μια διετία. Θα πρέπει να αναλύσουμε την ε, κατάσταση στην πράξη, να δούμε τα υπέρ και τα κατά μετά την εφαρμογή του συστήματος και λόγω της οικονομικής κρίσης θα πρέπει να μην συμπεριλάβουμε στοιχεία που μπορεί να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις εταιρείε και στα κράτη-μέλη και τα εισοδήματά τους. Θα πρέπει λοιπόν να αγωνιστούμε κατά της φορολογικής και δημοσιονομικής κρίσης. Είναι σημαντικό τα κράτη-μέλη να διεξαγάγουν Μελέτε αντικτύπου δεν μπορούν ε, να εργαστούν στο κενό. Ε, βέβαια αυτό είναι και δική μα ευθύνη. Προφανώς ε, εδώ δεν θα συμφωνήσω πολύ με τον εισηγητή. Τώρα για άλλα ζητήματα φορολογίας θα πρέπει να εναρμονίσουμε το, το σύστημα τιμολόγησης αλλά να ακολουθήσουμε και την αρχή της επικουρικότητας. Δηλαδή προφανώς δεν θα πρέπει να δεχτούμε τροποποιήσεις που θα αυξήσουν το κόστος για τις ε, εφορίες, της φορολογικής αρχής. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να πω ότι κατά την άποψή μου η κοινή ενωπημένη φορολογική βάση δεν θα πρέπει να βασίζεται στο παράγοντα του εισοδήματο και των πωλήσεων. Ε, μια παράμετρο πολύ δύσκολο να την αποτιμήσουμε. Θα συμφωνήσω λοιπόν εδώ με τον εισηγητή. Αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τον αριθμό εργαζομένων. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το στο οποίο να βασιστούμε. Και το φόρουμ είναι μια πολύ καλή ιδέα, διότι εκεί θα πρέπει να υπάρχει μια εντολή για εξοδικαστικές ε, επιλύσεις διαφορών, καθώς και εξέταση προδικαστικών ε, ερωτημάτων που μετά μπορεί να απευθυνθούν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να επιληφθούν τα δικαστικά συστήματα των δικατομελών. Οι δικαστές είναι οι μόνε αμερόληπτες αρχές που θα μπορούν να αποφαίνονται για τι διάφορε υποθέσει. Επίση, πολύ προσεκτικά πρέπει να εξετάσουμε το ζήτημα της αρμοδιότητας των αρμοδιοτήτων και της δικαιοδοσίας. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τις ενδεχόμενε συνέπειες και να παρατείνουμε τη χρονική περίοδο. Η κοινή ενοποιημένη φορολογική βάση δεν θα πρέπει να αποτελέσει ένα πλεονέκτημα κατά των ε, εθνικών συστημάτων ή κατά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Θα συμφωνήσω λοιπόν εδώ με τον εισηγητή και επίσης πιστεύω ότι θα πρέπει να παραμείνουμε πιστοί στις αρμοδιότητες που μας έχουν ανατεθεί, τις αρμοδιότητες δηλαδή της Επιτροπής μας, διότι η καθήλυνα αρμόδια Επιτροπή είναι η Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων. Σωστά επίση προτείνεται μετά από πενταετία να αποτιμηθεί κατά πόσον αυτό το προαιρετικό σύστημα να αποτελέσει ένα ενιαίο υποχρεωτικό σύστημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, περιμένω λοιπόν τη συνεργασία μα με τον εισηγητή και του υπόλοιπου σκιώδει για να καταλήξουμε σε ένα επιτυχέ αποτέλεσμα. Merci. Ευχαριστώ λοιπόν. Μήπω κάποιοι άλλοι θα επιθυμούσαν να πάρουν το λόγο, η κυρία Λεγκρίπ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε πολύ σύντομα, αποφεύγοντας λεπτομέρειες τεχνικές σε σχέση με την πρόταση της Επιτροπής και αυτά που μας προτείνει ο συγητής μας, θα ήθελα να επιμείνω στη σημασία αυτού εδώ του θέματος, η πολιτική του διάσταση και φυσικά τα θέμα που έχει να κάνει με την φορολογική πτυχή εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα διακύβημα πολιτικής φύσεως, πολύ συγκεκριμένο, πολύ δυνατό, έχει να κάνει με την, θα λέγαμε, με μια ενοποίηση της φορολογικής πολιτικής, θα χρειαστεί μεγαλύτερη σύγκληση οικονομική ε, από όλες τις χώρες μέλη. Και είναι αυτό μια απαραίτητη ε, συνθήκη για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε και τον νομισματικό μας πυλώνα εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή χρειάζεται μια ενισχυμένη φορολογική ε, προσέγγιση. Ακούμε ότι η Επιτροπή δεν έχει προχωρήσει τόσο δυνατά, τόσο, δεν έχει πάει τόσο μακριά. Αλλά θα πρέπει να προσχωρήσουμε ότι το, το, το καλύτερο μπορεί να είναι εχθρός του καλού. Θα πρέπει να προχωρήσουμε πάνω στη βάση που έχουμε και θα, αν το πετύχουμε αυτό θα έχουμε προ... ήδη μια επιτυχία. Είναι σημαντικό λοιπόν να διηγηθούμε προς τη σύγκληση. Αυτό είναι το οποίο επιθυμούμε. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, άλλες παρεμβάσεις. Όχι. Λοιπόν, θα δώσω το λόγο στην Επιτροπή. Υπήρξαν πολλά αιτήματα για μια παρέμβαση της Επιτροπής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε ιδιαίτερος για τι προτάσεις επί τη έκθεση, Βλέπουμε ότι κάποιες από αυτές είναι πολιτικού χαρακτήρα, αλλά υπάρχουν και τροπολογίε που απαιτούν ενδελεχή νομική ανάλυση. Ιδίω ό,τι αφορά το φόρουμ και το δικαίωμα υποβολή ερωτημάτων προ το Δικαστήριο του Λουξεμβούργου. Θα πρέπει λοιπόν να τα δούμε όλα αυτά κατά Τώρα, σε ό,τι αφορά κάποιε από τι παρατηρήσει, κατά πρώτον φαίνεται ότι το σύστημα ε, θα είναι προαιρετικό, προαιρετικό για τις εταιρείε των 100 μελών. Όμως αν ένα 100 μέλος ε, πει ότι δεν θέλει δύο συστήματα να λειτουργούν ταυτόχρονα, εκείνο θα αποφασίζει κατά πόσον θα εναρμονίσει ή θα ευθυγραμμίσει το δικό του εγχώριο σύστημα με τους κανόνες της ΚΕΘΕ οι οποίοι ούτως ή άλλως ε, αρχικά θα βασίζονται σε εθνικά νομοθετήματα όπως τα γνωρίζουμε είναι πολύ κοντά σε πολλά ε, συστήματα εθνικών ε, κανόνων, όπως τα γνωρίζουμε από τα κράτη-μέλη. Οι πωλήσει προορισμό είναι ένας παράγοντας που έχει χρησιμοποιηθεί στην ε, υπάρχουσα φόρμουλα, ώστε να προταθούν εισοδήματα στα κράτη-μέλη που δεν παράγουν αλλά των οποίων οι καταναλωτές καταναλώνουν προϊόντα και υπηρεσίες διαφορετικών ευρωπαϊκών εταιριών. Εάν λοιπόν αφαιρέσουμε αυτό τον παράγοντα των πωλήσεων των πωλήσεων ένα προορισμό, θα δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στα φορολογικά εισοδήματα, αυτά καθεαυτά, για κάτι μέλη τα οποία δεν έχουν περιουσιακά στοιχεία ή έχουν εργαζομένους που παράγουν τις, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Αυτό αλλάζει την κατανομή των φορολογικών εισοδημάτων μεταξύ των κρατών εφόσον οι πωλήσει προορισμό ή οι πωλήσει μόνε του δεν χρησιμοποιηθούν ω κριτήριο. Θα πρέπει λοιπόν να το εξετάσουμε για να δούμε πώ μπορεί να ληφθεί υπόψη. Think, ε, Νομίζω αυτά είναι τα σημαντικότερα σχόλια που είχα να κάνω. Ευχαριστώ. Merci. Ευχαριστώ. Θα ξαναδώσω τώρα το λόγο στον εισηγητή. Μια ερώτηση μόνο. Μια και έχω το λόγο και δεν είμαστε και πολύ παρόντες, έχουμε χρόνο. Εξή ερώτηση. Ε, ε, έχοντας μια ελάχιστη, ένα εναρμόνιση και λαμβάνοντας υπόψη το διάλογο σήμερα, δεν φοβάται ότι μπορεί κανείς να ενισχύσει τις ανισότητες και τις δυσκολότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για κάποιες χώρες μέλη. Αν κανείς δεν πάρει τις διατάξεις οι οποίες για μένα τουλάχιστον μου φαίνονται επιτακτικές. Πάμε προς τη σωστή κατεύθυνση λοιπόν ή μήπω ε, ενισχύουμε τις ανισότητες που υπάρχουν, ε, διευρύνουμε το πρόβλημα. Well, Ευχαριστώ. Ασχολούμαι με τα ζητήματα της πολιτικής κάμποσα χρόνια. Βεβαίω. Καλό είναι να έχει κανεί στόχο τα ουράνια, αλλά αυτό δεν πετυχαίνει πάντοτε. Κάποιες φορές πρέπει να είναι και πιο πραγματιστής και προσγειωμένος. Εάν θέλετε, όπως είπε η κυρία από την Επιτροπή, να πετύχει κάτι. Έτσι λοιπόν, Καταλαβαίνω τα επιχειρήματά σας υπέρ της εναρμόνισης. Αλλά από τη δική μου την άποψη, το άλλο ζήτημα που θα πρέπει να μας απασχολήσει είναι η νομιμότητα. Είναι πολλά αυτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση που σήμερα συμβαίνουν με έναν τρόπο πλήρως αδιαφανή. Καμιά δημόσια συζήτηση. Τα κράτη-μέλη και οι πολίτες τους δεν εμπλέκονται ιδιαίτερως αυτό είναι ένα ζήτημα κρίσιμης σημασίας και όχι μόνο οικονομικής αλλά και πολιτικής. Η περίοδος είναι κρίσιμη γενικότερα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ προέρχομαι από μια χώρα που όπως μάλλον θα γνωρίζετε πάντοτε ζούσε με υψηλούς φόρους. Δεν είχαμε πρόβλημα. Τους έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια, εντάξει, αλλά έχουμε συνηθίσει. Έχω συνηθίσει σε αυτή την ιδέα και στην ιδέα ότι οι πολιτικοί που προβλέπουν τους υψηλούς φόρους θα έπρεπε να μπορούν να, βγουν στο δρόμο και να μπορεί κανείς να συζητήσει μαζί τους σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Γνωρίζουμε ότι το κοινοβούλιο αυτό νομίζω κατά 45% προέβλεψε μάλλον ένα κύκλο εργασιών από τα φορολογικά 45% και ένα 25% από άλλες χώρες. Αυτό έχει να κάνει με την κυριότητα των ε, ίδιων των χωρών. Δεν λέω να μην λάβουμε δραστικές αποφάσεις, κάνει μια αντίρρηση. Όμως να σκεφτούμε και ότι δεν πρέπει να δαγκώσουμε με πολύ δύναμη. Θα δούμε πού θα καταλήξει όλο αυτό. Γνωρίζω ότι η κυρία Τίσεν ε, στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων προτείνει λίγο πολύ να ακολουθήσουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκή Επιτροπής. Δεν αλλάζει σχεδόν τίποτε. Αυτό είναι το σκηνικό. Ε, επίσης για την ερώτηση του κυρίου Ντεγιόνγκ. Ξέρω ποιες είναι οι απόψεις Όμως η επικουρικότητα, όπως έλεγε και η κυρία Ρόιτοβα, πρέπει να ληφθεί υπόψη. Και από τη δική σας την άποψη, κύριε, Δεν αρκεί να πούμε αυτό θα πρέπει να κάνουμε τώρα και με οποιοδήποτε κόστος να το πράξουμε. Όχι. Πρέπει να τα σκεφτούμε και αυτά. Ίσως με την ενδεχόμενη τροποποίηση της συνθήκη, να μπορούσαμε και αυτό να το λάβουμε υπόψη. Ίσως λέω. Από τη δική μου λοιπόν την σκοπιά στηρίζω την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και γιατί τώρα προτείνω την αλλαγή στην, στον αναδιανεμητικό χαρακτήρα του συστήματος με τον παράγοντα των πωλήσεων είναι θέμα ισορροπίας. Αλλά όπως επίσης μάλλον γνωρίζετε, είναι και ένα από τα βασικότερα προβλήματα των μικρών χωρών, προκειμένου να δεχθούν την πρόταση. Εάν προσπαθήσουμε να υπολογίσουμε, δύσκολο βέβαια, αλλά αν προσπαθήσουμε να υπολογίσουμε τι συμβαίνει, αυτό θα ωφελήσει κυρίως τις μικρές χώρες Συμφωνώ λοιπόν ότι χρειάζονται και άλλες αναλύσεις, μελέτες αντικτύπου, αλλά αυτό είναι μια απλή άποψη. Το όλο ζήτημα είναι περίπλοκο και μπορεί να μας παραπλανήσει. Όμως καλό θα ήταν να τα σκεφτεί όλα αυτά η Επιτροπή και με μια πιο προσεκτική ανάλυση να επανέλθει στην Επιτροπή μας. Αυτό νομίζω θα ωφελήσει την εξέταση του όλου ζητήματος. Ολοκληρώνοντας, να πω ότι θα μπορούσα να δεχτώ οι δραστικές και ριζοσπαστικέ αλλαγές να μην παραμείνουν, αλλά δυσκολεύομαι ιδιαίτερος να δεχτώ το σύστημα να είναι υποχρεωτικό και να υπάρχει ελάχιστος φορολογικός δείκτης. Και αυτό γιατί έχω ακούσει εκπροσώπου του χώρου. Δεν θεωρώ ότι αυτό είναι αθέμητο. Εκείνοι δημιουργούν τι τέσσερι εργασία. Χρειαζόμαστε λοιπόν περισσότερες ανταγωνιστικές εταιρείε στην Ευρώπη. Εάν δεχτούν ένα τέτοιο σύστημα, θα πρέπει τουλάχιστον αυτό να προβλέπει μια μεταβατική περίοδο. Να τους ακούσουμε νομίζω λοιπόν. Για μένα αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ζω σε μια χώρα όπου έχουμε εγώ και κυρία Μπίλτ τέλο πάντων έχουμε πολύ ψηλού φόρους. Ίσως περισσότερο από κάθε άλλον σε αυτή την αίθουσα. Τους αντέχουμε λοιπόν τους ψηλούς φόρους, αλλά θα πρέπει να είναι στοχευμένοι και αποτελεσματικοί και να αποφασίζονται και σε εθνικό επίπεδο, όπως ως τώρα. Sí. Καλώς. Η κυρία Ρόιτεβα ξαναζήτησε το λόγο και αφού έχουμε το χρόνο, ο κύριος Τζογιούγκ θέλουν να ξαναπάνουν το λόγο και υπάρχει δυνατότητα λοιπόν να δώσω το λόγο στην κυρία Ρόιτεβα. Ευχαριστώ. Το θέμα της νομιμότητας που έθιξε ο συνάδελφος, η Επιτροπή μας και το Κοινοβούλιο γενικότερα, προφανώς πρέπει να έχουμε υπόψη ότι έχει αναλάβει να οικοδομήσει την ενιαία αγορά. Για κάθε εταιρεία με διασυνοριακή λειτουργία, είτε είναι μικρή είτε μεσαία, θα αντιμετωπίσει πρόβλημα εάν έχουν δραστηριότητα εκτός συνόρων, η φορολογική τους βάση θα υπολογίζεται διαφορετικά. Θα είναι λοιπόν ε, καθοριστική σημασία η απόφαση αυτή. Αυτά από τη σκοπιά της εσωτερικής αγοράς. Τώρα, ε, πολιτικές ε, παρατηρήσεις. Για όσους δεν θέλουν μεγαλύτερη ολοκλήρωση, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Εάν ενοποιήσουμε τη φορολογική βάση, Και εάν υπάρξει πολιτική βούληση, που τώρα δεν βλέπω να υπάρχει, τότε στο μέλλον αναγκαστικά θα εναρμονίσουμε και τους φορολογικούς δείκτες. Αυτό θα έπρεπε λίγο να μας θέτει σε επιφυλακή. Από την άλλη, το να προδικάζουμε ότι η ενοποίηση της εσωτερικής αγοράς δεν θα πρέπει να αποτελεί στόχο, ότι είναι ένα ταμπού και αυτό είναι λάθος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε την πρότασή τη και νομίζω ότι θα πρέπει να την αποτιμήσουμε. Και βάσει του διεθνούς εμπορίου και βεβαίως της αρχής της επικουρικότητας. Ένα τέτοιο σύστημα θα πρέπει να είναι πρακτικό Εάν όμως το μόνο που μας απασχολεί είναι οι εθνικοί προϋπολογισμοί, το ζήτημα είναι κατά πόσο να επιτελούμε τα καθήκοντά μας ως πολιτική λειτουργή. Αυτό νομίζω το θέμα είναι ιδιαίτερα περίπλοκο και θα συζητηθεί διαμακρών στο Συμβούλιο. Πάντως, από το Ευρωκοινοβούλιο καλό θα ήταν να αποστείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα και να μην μπλοκαριστεί το θέμα αυτό στην Επιτροπή μα. Ευχαριστώ. Ε, έχουμε τη συνήθεια και, και έχουμε καλήσει συνεργασία και συνεργαζόμαστε τακτικά με τα εθνικά κοινοβουλία. Ε, είναι εξάλλου η συνθήκη της Σαβώνας σε αυτό το θέμα. Είναι λοιπόν και αυτό μια δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα τα οποία έχουμε μέσω της συνθήκης στα χέρια μας. Ο Λίμ έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ. Να μην ξαναρχίσουμε το διάλογο. Όλοι, οι εισηγητές, οι σιώδεις εισηγητές έχουν ε, εκφραστεί. Εγώ να πω μια, κάνω μια παρατήρηση μόνο. Μπορούσε κανείς ε, σε αυτή τη σουρεαλιστική ένωση να προτείνει διάφορα πράγματα. Όποιος θέλει ας πούμε να πληρώνει φόρους τη στιγμή που συναντώμε τώρα μια πραγματικότητα όπου θέλει κανείς με θέματα ε, δημοσιονομικής να εφαρμόσει ποινέ, θα ήθελα να πω ότι ε, αυτό που συναντάμε σε, αυτή τη διαδικασία είναι ότι ζητάει κανείς πάντοτε ε, να καταβάλουν και να κάνουν προσπάθεια και να πληρώσουν ας πούμε, το λογαριασμό πάντοτε οι ίδιοι και οι ίδιοι. Ευχαριστώ Πρόεδρος. Κάποιος άλλος που θέλει το λόγο. Ο κύριος Ντεγιόν. Ευχαριστώ και σύντομα, κυρία Πρόεδρε. Οι, οι προτάσεις που γίνονται με βρίσκουν σύμφωνο. Σίγουρα θα πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα. Στην, ε, στις κάτω χώρες έχουμε 1,67% του ΑΕΠ. Δηλαδή θα είναι η αρνητική επίπτωση, θα λέγαμε, η μείωση. Και λαμβάνοντας τα μέτρα που παίρνουμε θα μπορούμε να έχουμε και τις ποινές εκ μέρους της Μέρκελ. Εμείς θα ήθελα να πω ε, ότι δεν είμαστε κατά αυτό το μέτρο. Εμείς έχουμε ένα ελάχιστο επίπεδο και σύμφωνα με τη δική μας εμπειρία σίγουρα είμαστε πολύ θετικοί σε αυτή την προσπάθεια ενοποιημένης φορολογικής βάσης. Ε, απλώς θέλουμε να έχουμε χρόνο, πιο πολύ χρόνο, για να μπορέσουμε να κάνουμε κάποιες προτάσεις τροποπολιών και είναι σημαντικό αυτό να γίνει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Πρόεδρο, συμφωνώ μαζί σας. Θα ξαναμιλήσουμε για το χρονοδιάγραμμα. Ο κύριος έχει το λόγο. Χαίρομαι που φτάνω στο τέλος της συζήτησης. Δεν ε, μπορούσα να παρευρεθώ γιατί ήμουν πρόεδρος σε άλλη συνάντηση με τον συνονόματο του κυρίου Σμιτ, ο οποίος ε, μας ε, παρουσίασε μια ομιλία για την ε, καινοτομία. Λοιπόν, για τα ζητήματα που τώρα αντιμετωπίζουμε, είναι πολύ επίκαιρο το ζήτημα αυτό. Το όλο ζήτημα της ανάπτυξης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ορισμένες χώρες η φορολογική η φορολογία των εταιριών μάλλον και το τι γίνεται με τις πιστώσεις των εταιριών, το τι εισοδήματα ε, μπορούν να αποκομίσουν οι εταιρείε βάσει του φορολογικού συστήματος, όλα αυτά είναι καθοριστική σημασία. Το πραγματικό ερώτημα εδώ είναι εάν θα πρέπει να επιδιώξουμε την αρμόνιση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ή εάν οι χώρες θα λάβουν τι δικέ του αποφάσει, εισάγοντα περισσότερη καινοτομία στα συστήματά του και βάσει των αρχών τη ενιαία αγορά. Νομίζω ότι πρώτα απ' όλα επί αυτού πρέπει να συμφωνήσουμε. Και έπειτα, στα κράτη-μέλη γενικότερα, πρέπει να δούμε τι αρχέ, ε, την ελευθερία μάλλον του να ορίζουν μόνε του προλογικού του δείκτε. Ω τώρα, στα περισσότερα κράτη-μέλη, αυτό το θέμα είναι άμεσα συνδεδεμένο με την κυριαρχία τη κάθε εθνική χώρας. Οπότε, μετά τις συζητήσει των μελών της Ευρωζώνης, βλέπουμε οι αποφάσεις αυτές να είναι κρίσιμες. Τα κοινοβούλια βρίσκονται σε όλο ένα και πιο δυσάρεστη θέση. Εφόσον δεν μπορούν να σχεδιάσουν το φορολογικό σύστημα όπως θα έπρεπε. Ξέρετε τι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ της δικής μου χώρας και του κυρίου Σμιτ. Ε, είναι πολύ σοβαρές ε, οι διαφορές μεταξύ της παρακράτησης φόρων μεταξύ των δύο. και το τι γίνεται με το όλο σύστημα κοινωνικής προστασίας, κοινωνικών επιδομάτων και ούτω καθεξής. Και οι διαφορές συνεχίζονται μεταξύ των χωρών. Δεν νομίζω ότι τα κοινοβούλια ή οι χώρες ε, αναμένουν αναγκαστικά να οριστούν αυτή η τομή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το επιλύσουν τουλάχιστον οι χώρε μέλη τη Ευρωζώνη. Θα πρέπει, εφόσον υπάρξει ενοποιημένη φορολογική βάση για τι εταιρείε, αυτό να μην αποκλείσει άλλους ε, πολιτικούς τομείς που αφορούν την ε, οικονομική σύγκληση. Διότι αν αντιμετωπίσουμε μόνο έναν τμήμα του όλου ζητήματος που θα έπρεπε να τεθεί επιτάπητος, δεν θα προμελήσεις. Και επανέρχομαι στο αρχικό μου ερώτημα, εν κατακλείδη. Εάν οι χώρες που τα πάνε πολύ καλύτερα στη μεταφορά τεχνογνωσίας, στην έννοια νέων εταιριών και την καινοτομία, ε, σχετίζουν τις δραστηριότητες αυτές με το φορολογικό τους σύστημα και την οικονομική τους ανάπτυξη, αυτό θα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον ως δίδαγμα. Ίσως θα πρέπει να υπάρξει ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ χωρών που δεν τα καταφέρνουν τόσο καλά. Και οι χώρε να μπορούσαν να αποφασίσουν μόνε του εάν αυτό είναι κάτι συνετό που θα πρέπει να το πράξουν. Βεβαίω, έτσι θα είχαμε μία λύση που θα καθοριζόταν βάσει των αναγκών τη αγορά. Διότι οι περισσότερε εταιρείε θα μετακινούνταν σε μια χώρα που θα ε, του επιφύλασε καλύτερη φορολογική μεταχείριση σε αντίθεση με άλλε. Δεν ξέρω εάν ε, θα ήθελε ο εισηγητή να συμβεί κάτι τέτοιο, γιατί τότε θα, είχα, θα ήταν αυτό πολύ ευνοϊκό για μένα τον ίδιο. Δεν ξέρω αν θα ήταν έτοιμο να το στηρίξει. Sí. Bon, alors... νομίζω και όλοι όσοι εκφρασίγαν εδώ δείχνουν ότι είναι ένα πολύ περίπλοκο ε, θέμα. Έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα ε, πολύ αυστηρό, πιεστικό. Προβλέθηκε ε, προθεσμία κατάσταση τροπολογιών 8 Δεκεμβρίου και προτείνω να κάνουμε ό,τι κάναμε με το προηγούμενο θέμα. Να μεταφέρουμε την προθεσμία κατάσταση τροπολογιών στην επόμενη Τετάρτη 14 του μηνός αν συμφωνεί τώρα και ο εισηγητής, με εξέταση των τροπολογιών όπως έχει προβληθεί 9 Ιανουαρίου, ψηφοφορία στην ΙΜΚΟ 6 Φλεβάρι. Θα υπάρχουν εντωμεταξύ συναντήσεις ανάμεσα στον εισηγητή και στους χιώδη εισηγητές και η ψηφοφορία στην ΕΚΟΝ 29 Φεβρουαρίου με προβλεπόμενη ψηφοφορία στην Ολομέλεια τη 17η Απριλίου. Υπάρχει κάποια επιφύλαξη. Νομίζω ότι είναι ένα χρονοδιάγραμμα που είναι πολύ έτσι βολικό και μας επιτρέπει να δουλέψουμε σωστά. Δεν βλέπω κάποια αντίδραση. Έτσι λοιπόν φτάνουμε στο τέλος της ε, συνεδρίασίας μας. Κατά εξαίρεση πολύ νωρίτερα, κλείνουμε. Θα σας εύχομαι ε, καλή ξεκούραση ενώπιστον για τον εορτών. Ευχαριστούμε και τους διερμηνείς και ένα δωράκι μικρό γιατί συχνήθω σα τρώμε το χρόνο και δουλεύουμε λίγο περισσότερα. Τώρα λοιπόν καλή ξεκούραση και σε εσά, αλλά κλείνοντα θα δώσω το λόγο στον πρόεδρο μας. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ την Μπερνάντα Τιμπερνιό για την τόσο επιτυχή προεδρία, στην ε, συνεδρίαση, επιτυχή εταιρική σχέση επίση. Να πω ότι θα υπάρξει άλλη μια συνεδρίαση πριν τα Χριστούγεννα στι 20 Δεκεμβρίου. Στι 3 το μεσημέρι. Και καθώ θα κλείνει η Πολωνική Προεδρία, θα δούμε μια σειρά από θέματα. Επίση, να σα ενημερώσω δημοσίω Νομίζω δεν αποτελεί μυστικό ότι στις 20 Δεκεμβρίου θα είναι η τελευταία φορά που ο κύριος Ντάν θα είναι μαζί μας ε, στο Προεδρείο. Θα αλλάξει πόστο. Θα αναλάβει πολύ σημαντικότερα καθήκοντα. Είναι κάτι για το οποίο επισήμως δεν έχω ενημερωθεί, αλλά ο λόγος που σας το λέω αυτό είναι γιατί θα ήθελα να σας προσκαλέσω για ένα ποτό μετά τη συνεδρίαση της 20 Δεκεμβρίου. Η τελευταία συνάντησή μα με τον Ντάν. Θα το ευχηθούμε λοιπόν καλή τύχη στη νέα του θέση και θα δούμε τι θα γίνει με την αντικατάστασή του. Ε, ήθελα λοιπόν αυτό να το ανακοινώσω δημοσίω και θα τον ευχαριστήσω θερμά και τότε. Διότι υπήρξε επικεφαλή τη Γραμματεία από τότε που ξεκίνησε τι εργασίε τη το 2004. Ήταν μια νέα επιτροπή που συστήθηκε το 2004 και βεβαίω θα προσκαλέσω και τον προκατοχό μου, τον κύριο Μακάρθη, να, μας, ε, να έρθει μαζί μα, διότι Όπως ξέρετε μάλλον, δεν θα μπορέσω να τον προσκαλέσω γιατί τον χάσαμε πριν 5-6 χρόνια. Σας εύχομαι καλό βράδυ και ευχαριστώ και εγώ ιδιαίτερα στους διερμηνεί.